Okay. Dear colleagues, we can uh, start. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε. Πρώτο θέμα έγκριση της ημερήσιας διάταξης, αν δεν διαφωνείτε, το σχέδιο μπορεί να εγκριθεί χωρίς τροποποίησης. Ε, σημείο 2. Ανακοινώσεις. 2 Ιουνίου είχαμε προβλέψει συνεδρία της Επιτροπής μας, η οποία ματαιώθηκε. Έχουμε ε, ενημέρωση για μια αποστολή στο Λονδίνο, στο ΝΕΟΦ ε, και θα τα βρείτε εκεί που γνωρίζετε. 21 γλώσσες έχουμε σήμερα και ως συνήθως ε, ηλεκτρονικά έχετε πρόσβαση στα έγγραφα και η συνεδρίαση όσοι ήθιστε μεταδίδεται απευθείας στο διαδίκτυο. 3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων τη 23 η Φεβρουαρίου, 21η και 22 η Μαρτίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει μέχρι την, το τέλος συνεδρίασης θα θεωρηθούν εγκριθέντα τα πρακτικά. Λοιπόν, και τώρα προχωρούμε στο βασικό σημείο. Παρίσταται ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριος Μάρος Σεύσκοβιτς. Καλωσορίσατε θερμά στην Επιτροπή μας. Έχουμε ανταλλαγή απόψε, όπω γνωρίζετε, με τον Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Αρμόδιο για την Ενεργειακή Ένωση ω μέρο του διαρθρωμένου διαλόγου. Ε, ξέρετε ότι έχουμε ένα τέτοιο ετήσιο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα πλαίσια αυτά, περιμένουμε να ακούσουμε με χαρά τι γίνεται με την εφαρμογή του προγράμματος δράσης ε, για το 2016 ε, και τις προτεραιότητες σας επέκεινα. Μετά τη συμφωνία που έχουμε ε, στόχος της ανταλλαγής απόψεων είναι να δούμε πώς προχωράει ε, και η νομοθεσία για το 2030 για τα ενεργειακά τα διάφορα θέματα που μας απασχολούν και για τις μεταφορές, εκπομπές ρήπων κτλ. Η Επιτροπή μας και μετά τη Συμφωνία των Παρισίων παρακολουθεί πάρα πολύ στενά την υλοποίηση αυτού του πλαισίου για το 2030, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμορφούται με τις ε, υποχρεώσεις που ανέλαβε στη διάσκεψη των Παρισίων. Σας καλωσορίζω και πάλι κύριε Επίτροπο και σας δίνουμε στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Λαβία. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, έχετε απόλυτο δίκιο. Την τελευταία φορά που είχαμε ανταλλαγή απόψε ήταν ακριβώ πριν από ένα χρόνο, πολύ λίγο μετά την ε, υιοθέτηση τη ε, στρατηγική τη Ένωση για την Ενέργεια. Ένα χρόνο θα έλεγε κανεί ότι δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλο διάστημα, ειδικά όταν μιλάμε για τη χάραξη πολιτική, αλλά πιστεύω πω όλοι θα συμφωνείτε ότι από την ε, από την εισήγηση των προτάσεων για την ε, στρατηγική περινέργεια της Ένωσης έχουμε προχωρήσει πολύ. Ξεκινήσαμε με την εφαρμογή, ε, συνεργαστήκαμε ώστε να είναι επιτυχής η σύσκεψη των Παρισίων και ορισμένοι από εσά μάλιστα ε, συνεργαστήκατε για τα διάφορα εργαλεία για την Ένωση, την ενεργειακή. Και νομίζω πως όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά γιατί το να μπορέσουμε να έχουμε την Ενεργειακή Ένωση ως κοινό σχέδιο, κοινό όραμα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και να επιτύχουμε σε αυτήν την προσπάθεια σημαίνει κινητοποίηση της κοινή γνώμης για να το στηρίξει αυτό το σχέδιο. Δηλαδή η παρουσίαση του προγράμματος και εκστρατεία στα κρατημέλη ώστε να εξηγήσουμε γιατί πρέπει να υπάρξει μετάβαση ε, κατεπηγόντων στην κοινωνία του χαμηλού, χαμηλής καταναλωσάνθρακα. Όσοι και μεταβήκατε και εσείς στα κάτι μέλη, θα φαντάζομαι θα συμφωνείτε μαζί, σας, μαζί μου ότι ήταν εντυπωσιακό ο ενθουσιασμός που επικρατεί σε ολόκληρη την Ένωση όταν είχαμε επαφές με τα κοινοβούλια, με τους βουλευτές, ε, με τους, ε, την κοινωνία των πολιτών, με τους πολίτες, ε, με τους επιχειρηματίες και τα πιο σημαντικά ερωτήματα δεν ήταν το γιατί, αλλά το πώς, πότε και πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε αυτά τα project. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι έγινε μια καλή αρχή, υπήρχε μια ισχυρή αίσθηση δέσμευσης και οικειοποίησης του project αυτού από το Ευρωπαϊκό Κοινό. Επόμενη πολύ σημαντική εξέλιξη από την τελευταία μας συνάντηση ήταν ε, το, η εκδήλωση στην οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος, δηλαδή η COP21 που κατέληξε στη Συμφωνία των Παρισίων και είμαι υπερήφανος που την υπέγραψα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τέσσερις εβδομάδες στη Νέα Υόρκη. Και όλοι όσοι συμμετείχαμε ήμασταν υπερήφανοι γιατί σπάσαμε το ρεκόρ των χωρών που υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία σε μια μέρα, σε μια τέτοια συμφωνία μάλλον σε μια μέρα. Πραγματικά πρόκειται για μια παγκόσμια κινητοποίηση. Γιατί είναι σημαντικό τώρα αυτό για μας τους Ευρωπαίους. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η συμφωνία να μας δώσει μια σαφή κατεύθυνση ε, προς ε, τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε. Με αυτά τα δύο παραδείγματα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι ε, για το project αυτό πραγματικά βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή θέση, καλή φάση και σήμερα θέλω μαζί σας να δούμε πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε και να συνεργαστούμε καλύτερα για ώστε να έχουμε βιώσιμο μέλλον. Για να τα καταφέρουμε αυτά, αυτό, τρία στοιχεία του, του τριγώνου βιωσιμότητας θα πρέπει να εφαρμοστούν και να αλληλοενισχύονται. Πρώτον, καλή πολιτική. Δεύτερον, βιώσιμη χρηματοδότηση. Και βέβαια, τεχνολογία ε, υψηλής ποιότητας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αναλύσω τις τρεις γωνίες αυτού του τριγώνου. Πρώτον, η πολιτική. Έχουμε ε, λοιπόν διάφορα αλληλένδετα πακέτα και ξέρω πως είχατε ανταλλαγή απόψεων με τον συνάδελφο Αρία Κανιέτε που ήδη έχει αρχίσει να παρουσιάζει αυτά τα πακέτα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι σύντομο ω προ αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει πριν το καλοκαίρι είναι να ε, να συγκλίνουμε στους στόχους ε, για τα αέρια του θερμοκηπίου όπως συμφωνήθηκαν στο Παρίσι από τους αρχηγούς των κρατών και των κυβερνήσεων και να μετατραπούν αυτά και να ανατεθούν στα κρατημέλη στο πλαίσιο των εθνικών τους ευθυνών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διευκολύνει την κατάσταση, να δημιουργήσει ένα θετικό περιβάλλον και είμαι σίγουρο πως γνωρίζετε πως αυτή τη στιγμή έχουμε επαφές διαρκείς σε πολιτικό επίπεδο με τα κρατημέλη που εξηγούμε την προσέγγισή μας τη φιλοδοξία μας και τι θα χρειαστεί σε αυτή τη διαδικασία και βέβαια τις τεράστιες προσπάθειες που πρέπει να κάνει να καταβάλει κάθε ε, κράτος μέλος για αυτή την κοινή στο κοινό εγχείρημα. Στον τομέα των μεταφορών, για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερο ώστε να ενισχύσουμε την κινητικότητα χαμηλού άνθρακα, να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα και να μετακινηθούμε από τη χρήση ε, των παραδοσιακών ε, ορυκτών καυσίμων στη χρήση νέων καυσίμων για την χρήση νέων οχημάτων, νέων τεχνολογιών, καθώς και την ενσωμάτωση των συστημάτων ICT στις ε, μεταφορές. Μαζί θα έχουμε μια τέτοια τέτοια απόφαση, θα υιοθετήσουμε μια τέτοια απόφαση, σχετική απόφαση πριν τι ε, διακοπέ. Επίση, σημαντικό τομέα είναι ο τομέα των κτηρίων. Μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας περί ενεργειακής απόδοσης και αποδοτικότητας των κτηρίων που θα υποβληθεί αμέσω μετά τις καλοκαιρινέ διακοπέ. Θα πρέπει να αλλάξουμε το πω σκεφτόμαστε και ενεργούμε για τα κτίρια από την παραδοσιακή άποψη του, του, του παθητικού κτίριου σε μετακίνηση σε μια e e, ευφυή κατασκευή που είναι πιο αποτελεσματική, λειτουργεί με πιο αυτοματοποιημένο τρόπο και ίσω να είναι και σε θέση να ξαναφορτίσει τις μπαταρίες του στο υπόγειο. Ας σκεφτούμε δηλαδή ποιες δυνατότητες υπάρχουν, ποιες τεχνολογίες υπάρχουν, ώστε να καταστήσουμε τα κτίρια μας ε, συνδετικούς κρίκους, να τα κάνουμε συνδετικούς κρίκους ώστε να μπορέσουμε να, μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην οικονομία του 21ου αιώνα και στις ε, συνδεδεμένες υποδομές. Ε, πρόκειται βέβαια ε, και για στοιχεία τα οποία εδώ και χρόνια γνωρίζουμε ότι δηλαδή το μερίδιο του ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες θα περάσει στο 50% μέχρι το 2030 και γι' αυτό και πρέπει να αναμορφωθεί και η αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Νέα οδηγία για την, τις ανανεώσιμες καθώς και, η πρόταση για τη διακυβέρνηση θα παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να επιτύχουμε τους στόχους ανανεώσιμες, ανανεώσιμες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2025. Δεύτερο γωνία του τριγώνου είναι η ε, χρηματοδότηση. Η διθέσπιση στόχων, πολιτικών στόχων είναι σημαντική, αλλά δεν είναι αρκή θα πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση και επαρχή, επαρκής βιώσιμες επενδύσεις. Όπως γνωρίζετε, τα επίπεδα επενδύσεων δεν έχουν ακόμα επανέλθει στα κανονικά τους επίπεδα μετά την κρίση. Βλέπουμε και προβλέπουμε ε, ε, ε, ανάγκες 150 με 200 δις ευρώ μόνο και μόνο μέσα στο τομέα του ηλεκτρισμού μέχρι το 2030. Τεράστια πρόκληση που πρέπει να χειριστούμε σε πολλά μέτωπα. Τα διευθυντικά ταμεία και το ΕΦΣΙ είναι τα βασικά μέσα για να περάσουμε σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Και αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Το επενδυτικό πρόγραμμα Juncker έχει βοηθήσει στο να βρεθούν βιώσιμε πράσινε επενδύσει σε ολόκληρη την Ένωση για δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ένα μόνο χρόνο αυτό το ταμείο στηρίζει 64 projects με πάνω από 100 δισεκατομμύρια επενδύσει σε ολόκληρη την Ένωση. Και μάλιστα πάνω από το ίμιση αυτών των ε, projects που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής αφορούν ανανεώσιμες ενέργειες, επάρκεια στην ενέργεια και ενεργειακές επενδύσεις. Βεβαίως, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μόνο δεν μπορούμε να ενεργήσουμε, να γνωρίζουμε όλο και περισσότερο πως οι πόλεις παίζουν σημαντικό ρόλο και γι' αυτό δουλεύουμε για μια συγκεκριμένη ε, θηρίδα, one-stop shop για τις αστικές περιοχές και ξεκινάμε το Άμστερνταμ, ώστε να μπορέσουμε με αυτό το μέσο να συγκεντρώσουμε για πρώτη φορά όλα τα στοιχεία που αφορούν την κάθε πόλη, έτσι ώστε οι πόλεις πιο εύκολα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δυνητικές πηγές χρηματοδότησης. Αυτή η πλατφόρμα θα έχει σημαντική προσθέμενη εξήγηση για τοπικές αρχές, θα τους διευκολύνει να, να συμμετέχουν δραστήρια και να οικοδομούν βιώσιμες κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αφού συζητήσαμε την ατζέντα για τις ευφυεί πόλεις, στις διάφορα ταξίδια έχουμε ε, δει ότι υπάρχει επίδραση, υπάρχει επιρροή, ε, πρόκειται για πράγματα που μπορούν να αναπαραχθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχουμε 7.000 δημάρχους που συνυπέγραψαν το σύμφωνο των δημάρχων και το ενδιαφέρον αυξάνεται διαρκώς και σε όλες τις υπήρους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Αφρική, μια ήπειρο που επισκέφθηκα ως ε, μέρος ε, της εκστρατεία ε, συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίησης στην Προχωρώντας προς την COP21, είδαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουμε πολύ στενά, να συνεργαστούμε πολύ στενά με τους Αφρικανούς εταίρους μας, ώστε να μπορέσουν να οικοδομήσουν ε, δυνατότητες για να συνεργαστούμε μαζί σε κοινέ πλατφόρμες, να μοιραστούμε γνώσεις, ε, εμπειρίες και να μπορέσουμε να έχουμε και κατάλληλη χρηματοδότηση. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση με επικέφαλή τον ε, συνάδελφο Μίμητσα συμμετέχει στην Αφρικανική Πρωτοβουλία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας πολύ δραστήρια και συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να συνεργαστούμε με τους Αφρικάνους εταίρους για καλύτερη πρόσβαση στην ενέργεια. Τρίτο και τελευταίο στοιχείο του βιώσιμου τριγώνου που είναι η έρευνα, ε, τεχνολογική έρευνα και καινοτομία. Όλοι συμφωνούμε ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μια καινούρια βιομηχανική επανάσταση με καινοτόμο πνεύμα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ε, επισκεπτόμενος ε, πόλεις και περιφέρειες ε, βλέπουμε τα ίδια πράγματα και θα τα βλέπετε κι εσείς. Είμαι πεπισμένος πως οι Ευρωπαίοι όχι μόνο θα είναι κομμάτι αυτής της επανάστασης αλλά θα δώσουν, θα την προσανατολίσουν κιόλας και θα την σπρώξουν προς τα μπρος. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ένα μια στρατηγική, ολοκληρωμένη στρατηγική καινοτομία, έρευνα καινοτομία και ανταγωνιστικότητα που θα περιλαμβάνει τη βιομηχανία, τι ε, τηλεπικοινωνίε ε, και πολλού άλλου ε, τομεί, ενέργεια, περιβάλλον. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο χώρο έρευνα και τεχνολογία έτσι ώστε οι ευρωπαϊκέ βιομηχανίε να τοποθετηθούν στο σωστό σημείο τη αλυσίδα. Το Νοέμβριο θα παρουσιάσουμε αυτή τη στρατηγική. Βέβαια αυτή η στρατηγική θα πρέπει να είναι εξωστρεφή και να ε, ενισχύει την συνεργασία στα θέματα της έρευνας και της ε, καινοτομίας μαζί με τους ε, συναδέλφους θα συνεργαστούμε σε δύο εβδομάδες θα συναντηθούμε έτσι ώστε να συζητήσουμε αυτό ακριβώς το θέμα βέβαια θα μπορούσα να θίξω και άλλα πράγματα ε, για παράδειγμα την ε, ε, ευαισθητοποίηση των ε, πολιτών ή την, τα προσόντα τα οποία χρειάζεται το εργατικό δυναμικό για να περάσουμε στην νέα εποχή χαμηλού, χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε επαρκή και υγιή στέγαση. Τέλος, να μιλήσω για τη διακυβέρνηση της ενεργειακής πολιτικής τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι πολύ σημαντική. Μια ισχύ, ένας ισχυρός μηχανισμός διακυβέρνησης θα είναι πολύ σημαντικός για να εφαρμοστεί η Ενεργειακή Ένωση. Θα υποβάλουμε μέχρι το τέλος του χρόνου προτάσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξει, ε, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Πάντοτε επιμένω σε μια νομοθετική πρόταση έτσι ώστε ακριβώς το Κοινοβούλιο να μπορεί να παίξει ένα πλήρη και αποφασιστικό ρόλο. Σύμφωνα με τις αρχές της ε, καλής νομοθέτησης η πρόταση αυτή θα εξυγχρονίσει τις υποχρεώσεις που υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μείωση της γραφειοκρατίας και ταυτόχρονα τα εθνικά σχέδια ε, κλίματος και ενέργειας ε, θα ε, τεθούν σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όλες οι πτυχές της ενεργειακής στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. σταματάω λοιπόν εδώ, γιατί θέλω να ακούσω και τη δική σας νόμη και τις εξελίξη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ακούσω τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας και να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων σύμφωνα με τα θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν με ενδιαφέρει να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο, Κομισιόν και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θα βρούμε την ευκαιρία. Για παράδειγμα, όταν θα υποβάλουμε το δεύτερο κομμάτι της Ενεργειακής Ένωσης, το Δεκέμβριο δηλαδή του τρέχοντος έτους. Θα είναι και αυτό μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεχίσουμε το διάλογο μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με προσέξατε. Εγώ ευχαριστώ, ε, κύριε Αντιπρόεδρε. Αρχίζουμε το πρώτο γύρο των ομιλητών και δίνω αμέσω το λόγο στον Πέτερ Λίζα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και Αντιπρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφερθήκατε στη Συμφωνία των Παρισίων και την εφαρμογή της. Εκεί κυριαρχεί ένα βασικό στοιχείο που είναι το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Αλλά δεν θα πρέπει να μας απορροφήσει μόνο αυτό κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τα άλλα, με τον καταμερισμό των προσπαθειών και τα λοιπά για να ε, επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε για το κλίμα. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είμαστε κάπως επιφυλακτικοί ε, για κάποιες ενεργοβόρες ε, βιομηχανίες ε, το, οι 10 καλύτεροι παίρνουν 100% δωρεάν άδειες. Εμείς θέλουμε λίγο περισσότερες δωρεάν άδειες και πιστοποιητικά για να μην σηκωθούν να φύγουν οι βιομηχανίες. Στο έγγραφο θέσεων για το ΕΦΣΥ, για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, έχουμε κάνει και προτάσεις για το πώς μπορεί να διατηρηθεί ε, συνολικά, μάλλον για το ETS, ε, το θέμα ε, των ε, εκπομπών ε, και τι γίνεται με τις μεταφορές, τι γίνεται με την αεροπορία. Εγώ δεν μπορώ να πάω σε ένα εργάτη στη Χαλιβουργία και να του πω ότι μέχρι το 2030 πρέπει να έχει μειωθεί κατά 43% η εκπομπή της βιομηχανίας σου, ενώ στην αεροπορία είναι 10%. Ε, βέβαια αυτά πάντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός υπάρχει και ο ΑΕΚΑΟ και συζητούν αυτά τα θέματα να δούμε την έκβαση. Κάτι άλλο τώρα ε, που αναφέρθηκε στο έγγραφό σας για την Ενεργειακή Ένωση και το είχατε κάνει και σημαία, αλλά σήμερα δεν είπατε πάρα πολλά. Αυτή είναι η ενεργειακή απόδοση. Δηλαδή στην Ενεργειακή ε, Ένωση λέτε Energy Efficiency First. Εγώ διετέλεσα εισηγητή στο της Δότης Επιτροπής για την ε, εξέταση της οδηγίας για την έκθεση εφαρμογής και Κάναμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και σας παρακαλώ να τα διαβιβάσετε αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ληφθούν υπόψη τη πρότασή σας. Πρώτον, μέχρι τώρα η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση ισχύει μέχρι το 2020, εκπνέει μετά και συζητείται και σωστά αυτό το καιρό να παραταθεί η διάρκεια της μέχρι το 2030. Γιατί δεν το κάνουμε όπως γενικότερα στην κλιματική πολιτική και το εμπόριο εκπομπών ρήπων και μετά το 2030 θέλουμε να παραμείνει η ενεργειακή απόδοση. Και καλά θα ήταν οι επενδυτές να ξέρουν για να κανονίσουν την πορεία τους. Ας πούμε και το άρθρο 7 να διατηρηθεί και μετά το 2030 και να γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι αυτό το πρώτα η ενεργειακή απόδοση δεν ισχύει μέχρι το 20 αλλά ισχύει γενικώ. Για το στόχο επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Συμβούλιο μέχρι τώρα ε, αναφέρει 27% ότι είναι στόχος το ποσοστό στο Κοινοβούλιο. Ε, διαφωνούμε για το πόσε θα είναι οι οικονομίες, πάντως το 27% δεν ε, ανταποκρίνεται στο σύνθημά μας πρώτα η ενεργειακή απόδοση και υπάρχουν και εκπτώσεις. που διώχνουν τις επενδύσεις δεν είναι καθόλου ρεαλιστικά. Στη μελέτη αντεκτή που παρακαλώ να προσγειωθείτε λίγο και πραγματικά να είναι πρώτα η ενεργειακή απόδοση και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ματία Γκρότε, από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αγαπητέ Μάρο, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε σχέση με αυτό το τρίγωνο, καλή πολιτική, καλή χρηματοδότηση και καλή τεχνολογία. Είναι τρίγωνο αυτό. Την περασμένη εβδομάδα έγινε κάποιος άλλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ενεργειακή πολιτική, έβγαλε μια ανακοίνωση κομισιών για το θέμα των μήνυ ε, φορτηγών. Αυτό είναι ε, μάλλον το, το, το μήνυ πυρηνικών σταθμών. 30 χρόνια μετά το Τσερνομπίλ ε, και τη Φουκουσίμα, δεν νομίζω ότι η ενεργειακή πολιτική στο μέλλον είναι η ατομική ενέργεια και η πυρηνική ενέργεια. Ούτε μπορεί να λύσει τα προβλήματά μας. Και λένε οι συνθήκε και καλά κάνουν ότι για το ενεργειακό μείγμα αρμόδια είναι τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, στο μέλλον λίγη προσοχή όταν βγάζετε τέτοιε ανακοινώσει, γιατί δημιουργούν θόρυβο ω άλλο και μετά τρέχουμε να τα μαζέπουμε. Εγώ θα ήθελα και περισσότερε προδιαγραφέ, ιδιαίτερα στην κινητικότητα και σε άλλου τομεί. Θα πρέπει να κάνουμε τεράστιο βήμα προ τα εμπρό. Α πούμε, για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Πολύ ωραίο, μπορεί να γίνει με ανανεώσιμες αλλά μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν έχουμε δυνατότητα να φορτίζει το αυτοκίνητό του ένας Ευρωπαίος ας πούμε. Και είναι και πανάκριβο. Και θα πρέπει να έχει, ε, δεν υπάρχουν ενιαίες προδιαγραφές. Αν θέλει να διασχίσει την Ευρώπη με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, παίρνει ένα σωρό κάρτες μαζί του ε, για να μπορεί να πληρώνει την ενέργεια. Άλλο θέμα, μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Νομίζω ότι κάτι θα κάνουμε εκεί. Ε, είναι η έκθεση του Ιβο Μπελέτ για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Ε, θα ήθελα όμως, όπως είπε και ο Λίζε, να θυμίσω ότι αυτό ήταν πάγιο αίτημα και της Επιτροπής μας και στο Παρίσι να συνεισφέρει και η αεροπορία, η ενάρεια κυκλοφορία σε αυτό. Πώ να πα να το πει στη χημική βιομηχανία, σε άλλους κλάδους της βιομηχανίας, όταν συζητάμε με συνδικαλιστές πρέπει να τους εξηγούμε ότι η αεροπορία εξαιρείται, ξέρετε. Γιατί έχουν ιστορικές εξαιρέσει και παρεκκλήσει. Δεν γίνεται αλλιώ και φυσικά γίνεται και αλλιώ. Ε, και θέλω ε, λίγο περισσότερη πίεση από πλευρά. Άρα, μην σα ενοχλώ αφού μιλάτε και στο τηλέφωνο. Ε, να πιέσει, λέω, η Ευρωπαϊκή Επίτροπη και διεθνώς να συμφωνήσουμε. Και ακριβώς για τους τομείς που δεν ε, έχουν ενταχθεί το σύστημα εμπορία εκπομπών. Αυτό το effort sharing, ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων και των προσπαθειών θα πρέπει να γίνει στο εσωτερικό των 28 κρατών μελών. Liberal Group, uh, από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε Σεύκοβιτ για την συμβολή σας σήμερα. Εκατομμύρια ερωτήσει έρχονται στο μυαλό μου με τόσο ευρύ χαρτοφυλάκιο που έχετε. Είναι δύσκολο κανεί να εστιάσει σε ένα θέμα. Και επίσης ε, πολλά προβλέπονται μέσα στο δικό σας τομέα τους επόμενους μήνες, γιατί θα προσπαθήσω όσο γίνεται να εστιάσω σε κάποια πράγματα. Καταρχά, βεβαίως είχαμε πολύ επιτυχή συμφωνία των Παρισίων, αλλά έκτοτε βλέπω πολλά κράτη-μέλη που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις υποχρεώσεις που εμείς οι ίδιοι θεσπίσαμε για τους εαυτούς μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω δηλαδή επιστολές από διάφορα κράτη-μέλη που λένε στην Κομισιόν και σε άλλους ότι τα δέντρα τους, τα δάση τους είναι τόσο τεράστιοι δέκτες ε, λεκάνες ε, άνθρακα που θα πρέπει να εξαιρεθούν από τα μέτρα. Τους βλέπω να ζητούν ε, να εξαιρεθεί η δασοκομεία από την απόφαση για την κοινή προσπάθεια. Μιλούν για το γεωργικό τόμα και την εξαίρεση του, γιατί πρέπει λέει, να αναπτυχθεί, γιατί οικονομικά είναι εξαιρετικά σημαντικός και ούτω καθεξής. Για να είμαι λοιπόν ειλικρινής, βλέπω περισσότερες ε, κινήσεις προς περισσότερες εκπομπές από ότι προς λιγότερες. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο κατά τη γνώμη μου η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, συγκεκριμενοποιήσει το μονοπάτι που θέλει να ακολουθήσει προς την μείωση του άνθρακα προς το μέσα του αιώνα, μέχρι τα μέσα του αιώνα. Έχουμε φτάσει σε συμπεράσματα για τους στόχους του 2030. Χρειάζεται ωστόσο πάλι να θεσπίσουμε νέους ευρωπαϊκούς στόχους για την επάρκεια σε ενέργεια και περιμένουμε με ανυπομονησία τις προτάσεις σας. Βλέπουμε και γνωρίζουμε ότι το 2050 ότι μέχρι το 2050 μάλλον πρέπει να εκπέμπουμε 85%, λιγότερο ως ε, έως 95% λιγότερο ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε κάποια στρατηγική για μηδενικές εκπομπές και αυτή είναι συμβατή με τους στόχους που έχουν τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού και θα θέσετε κάποιους ενδιάμεσους στόχους γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να ενθαρρυνθούν περισσότερο ότι προχωρούν σωστά και ότι προσπαθούν όντως ε, και το να προσπαθούν να ξεφύγουν ε, ε, δεν είναι η σωστή στάση. Το άλλο για τα βιοκαύσιμα, η άλλη μου ερώτηση για τα βιοκαύσιμα. Αρκετά ξεκάθαρα μιλήσατε στην περσινή ακρόαση που κάναμε. Και στο θέμα, Λούκου, ήταν σαφές ότι δεν θα στηρίζαμε πια τα βιοκαύσιμα πρώτης γενναίας. Η ερώτησή μου είναι ποια είναι η θέση σας τώρα. Εξακολουθείτε να στηρίζετε την ίδια θέση, ότι δηλαδή τα βιοκαύσιμα της πρώτης γενιάς δεν είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Ούτε για το τομέα των μεταφορών, ούτε για το τομέα της αεροπλοείας. Γιατί επισκέφθηκα την ΙΚΑΟ στο αλλά πριν από δύο εβδομάδες και φαίνεται ότι μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στο στην αποκατάσταση, στην μάλλον στην ε, αντιστάθμιση των επιπτώσεων των βιοκαυσίμων και της πρώτης γενιάς δηλαδή βιοκαυσίμων. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η θέση της Κομισιόν για τα πρώτης γενιάς βιοκαύσιμα. Γι' αυτό θέλω να ξέρω ποια είναι η ισχύουσα άποψή σας για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Γκουε Κατερίνα Κονέτσνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, Ευχαριστούμε πολύ που προσπαθήσατε, που προσπαθείτε πάντοτε να μας κρατάτε ενήμερους σε ό,τι αφορά την Ενεργειακή Ένωση και γενικότερα το θέμα της αρμοδιότητάς σας. Ε, θα μιλήσω για κάτι το οποίο δεν σχολιάσατε. Η Κομισιόν είχε υποχρέωση στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης ε, να υποβάλει μια πρωτοβουλία σχετική με το οικονομικό πακέτο που αντίθετα με τα προηγούμενα δεν το, έχουμε, προσέξει επαρκώς σε ό,τι αφορά την καύση. Τι γίνεται με την καύση των αποβλήτων και, το, και την πρόταση που ήταν να υποβάλλεται. Η καύση είναι μια εναλλακτική λύση η οποία πιστεύω είναι πολύ χρήσιμη στον ενεργειακό τομέα. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας. Μερικές φορές η καύση όταν δεν γίνεται σωστά είναι χειρότερη από την αποθήκευση ή ε, ε, την ε, χρήση χιτά. Θα πρέπει η καύση να γίνεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με χαμηλές εκπομπές, πλην όμως σήμερα ε, αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε και προφανώς βλάπτει το περιβάλλον. Ε, έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις για την, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση τέτοιων και την χρήση τέτοιων εγκαταστάσεων. Ποια είναι η θέση σας για αυτό το θέμα σχετικά με την καύση. Μας είχατε μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία πέρσι. Πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα της κυκλικής οικονομίας και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Ευχαριστώ. Thank you very much. We have no members. Ευχαριστώ πολύ. Από τους Πρασίνους δεν έχουμε κανέναν. Η FTT ούτε. Θα δώσω μέσα στο λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει, κύριο Αντιπρόεδρος, για τον πρώτο αυτό γύρο. Thank you very much, Mr. Mr. Chairman. The first... Uh, Ευχαριστώ. πρώτη ότι ήταν από τον κύριο Λίζε. Χρήσιμες καταρχήν και μετά συμπληρώθηκαν και από τον κύριο Ματίας Γκρότε. Είναι γεγονό ότι η πραγματική εικόνα σήμερα είναι ότι μετά τη συμφωνία του, των Παρισίων και το, την ορμή που έδωσε ε, και πράγματι αυτή η συμφωνία ήταν ιστορικό επιτεύγμα. Βρισκόμαστε πλέον στη φάση που κάθε κράτος μέλος ε, με, μετράει, υπολογίζει τι σημαίνει για το ίδιο αυτή η συμφωνία. Οπότε τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή ε, ε προσπαθούν να προωθήσουν τις ιδιαιτερότητές τους στο καθένα. Ε, ε, ανάλογα με το που ταξιδεύει κανείς ε, ακούει διαφορετικά επιχειρήματα για τη βιομάζα στο βορρά και την σημασία της δασοκομείας και λοιπά, για παράδειγμα. Είναι σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας, διότι με αυτόν τον τρόπο διευκολυνόμαστε να καταλάβουμε και τα κράτη-μέλη διευκολύνονται να καταλάβουν τη θέση της αμοιβές θέσης. Είναι σαφές όμως ότι θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει επικεφαλής του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και η Συμφωνία του Παρισιού έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όχι μόνο υπέβαλε προτάσεις και ανέλαβε δεσμεύσεις, αλλά τη στήριξε αμέσως με νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες. Αυτή η συνεισφορά ήταν ιδιαίτερα σημαντική και θα συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών, για παράδειγμα, ε, ε, ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας σχετίζεται με αυτό που ονομάζουμε τα παρεπόμενα της Συμφωνίας των Παρισίων. Γεωργία, ενεργειακή αποδοτικότητα, αποδοτικότητα των ε, κτηρίων μας. Όλα αυτά σχετίζονται με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων. Μετά, το παιχνίδι έχει αλλάξει. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε αυτά που συνέβησαν όταν θέσαμε τους στόχους για το 2020, όπου ορισμένες από τις καινούργιες ε, χώρες ε, είχαν λάβει την άδεια να εκπέμψουν λίγο παραπάνω από ό,τι προβλεπόταν. Γιατί βρισκόντουσαν σε μια φάση βιομηχανικής ανάπτυξης. Τώρα πια όλοι πρέπει να κάνουν παρόμοιες προσπάθειες. Ε, αν θέλουμε να πετύχουμε το, τη μείωση 30% σε οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον, ε, στο σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών. Πρέπει να κάνουμε όλοι προσπάθειες και θέλουμε να πείσουμε τις κυβερνήσεις ότι αυτή η πρόταση, η πρόταση Κομισιόν είναι η πιο δίκαιη για κάθε κράτος μέλος. Πρέπει να το κάνουμε, διότι μόνο η συλλογική προσπάθεια θα μας επιτρέψει να πετύχουμε και να τηρήσουμε αυτούς τους ε, χρονικούς στόχους που έχουμε θέσει για το 2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τομέα της αεροπλοείας, Και εδώ είμαστε αυτοί που πιο πολύ επιμένουν και πιέζουν σε σχέση με τους διεθνείς παίκτες. Το σύστημά μας δουλεύει, μπορούμε να το αποδείξουμε τεχνικά. Καλύπτει τις εκπομπές ε, των αερίων θερμοκηπίου και είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να λειτουργήσει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως το πρόβλημα είναι ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι στην παγκόσμια σκηνή σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν σε συντονισμό με τα κράτη-μέλη προσπαθεί στο πλαίσιο του ΙΚΑΟ. Εγώ έχω συναντηθεί τελευταία με διάφορους παίκτες της, ε, του κλάδου και έχουν αντιληφθεί ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν. Το ξέρω αυτό, το καταλαβαίνω, το βλέπω. Θα πρέπει και η πολιτική αεροπορία να μειώσει τις εκπομπές Ελπίζω ότι μέχρι τον Οκτώβρη του φθήνοντος έτους ε, θα έχουμε πετύχει μια παγκόσμια συμφωνία για την εξουδετέρωση ε, της αύξησης των εκπομπών διεξουδίου του άνθρακα μέχρι το 2020. Το μηδενισμό της αύξησης δηλαδή. Δεν είναι πολύ υπερβολικά φιλόδοξο αυτός ο στόχος, μπορούμε να κάνουμε και παραπάνω. Αλλά από την άλλη μεριά ήδη θα ήταν μεγάλη επιτυχία αν ξεκινούσαμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον στόχο γιατί θα αποδείκνει ότι έχουμε μια παγκόσμια συμφωνία και θα μας βοηθούσε έστω και αυτή η επιτυχία ενός πρώτου ορόσημου η τηρήση μιας πρώτης προθεσμίας, έτσι ώστε να περάσουμε σε τα επόμενα βήματα. Το ίδιο ισχύει και με ένα άλλο κλάδο, τη διεθνή ναυσιπλοεία, ε, που για πολλά χρόνια διέφευγε της προσοχής μας, παρόλο που, είναι, που ρηπαίνει είναι σημαντικά. Και εδώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε παγκόσμια συμφωνία για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και τη συλλογή ε, συγκρίσιμων δεδομένων. Να δούμε ποιες είναι πιο ενεργειακά αποδοτικές ε, γραμμές, ε, με ποιο τρόπο επιτυχάνεται αυτό κλπ. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση, ε, θα εργαστούμε σε διάφορα επίπεδα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Καταρχήν πρέπει να αποκτήσουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για το ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι μας, ποιες οι φιλοδοξίες μας. Όπως γνωρίζετε, ε, ολοκληρώνουμε την μελέτη επιπτώσεων ε, αυτή την εποχή έτσι ώστε να ε, δούμε πώς πρέπει ακριβώς να δράσουμε έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους και για το 2030 και για την μετέπειτα εποχή. Στην Συμφωνία των Παρισίων αναλάβαμε την δέσμευση μείωσης των αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050 μεταξύ 80 και 90% και ε, η παγκόσμια οικονομία θα έπρεπε να είναι ουδέτερο πλευρά άνθρακα μέχρι το τέλος του αιώνα. Είμαστε λοιπόν σε στενή επαφή με τα κράτη-μέλη, διότι θέλουμε οι φιλοδοξίες μας ε, που θα παρουσιαστούν μέσω της οδηγίας ενεργειακής απόδοσης να περάσουν ε, και να μεταγραφούν με το σωστό τρόπο στα εθνικά σχέδια ενέργειας και κλίματος. και προσπαθούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη, εντατικά προσπαθούμε να τα πείσουμε ότι και αυτά θα πρέπει να κάνουν ό,τι τους αναλογεί. Τώρα, θα έχουμε με αυτόν τον τρόπο το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την τήρηση των επιτυχία των στόχων του 2030-2050, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να γίνει δουλειά και στα κράτη-μέλη. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να επεξεργαστεί ε, τα δικά του σχέδια, ενεργειακά και κλιματικά σχέδια σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Η ενεργειακή απόδοση θα παίξει σημαντικό ρόλο και ως τμήμα της διακυβέρνησης Ενεργικής Ένωσης ε, θα ε, υποβάλουμε, θα εκδώσουμε ε, ένα σκελετό για το πώς θα πρέπει, με τι θα πρέπει να μοιάζουν αυτά τα εθνικά σχέδια και θα περιλαμβάνουν ε, προτάσεις δράσεων για τη συμμόρφωση και με τους τρεις στόχους που έχουμε ε, θέσει. Για τις ενεργειακές πολιτικές και το έγγραφο το οποίο συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα, έγγραφο στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Χρότε, ε, αυτό αφορούσε την πρόταση εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς εμπειρογνώμονες της, ε, των κρατών μελών για, την, ε, για τις προτεραιότητες μας στις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας. Ε, κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τη λέξη πυρηνικός, πυρηνική, πυρηνικά, ξεσπάει η συζήτηση, το ξέρω αυτό. Θα ήθελα όμως να προσπαθήσουμε στο μέλλον όλοι μας ε, να εξασφαλίσουμε τη συζήτηση αυτού του θέματος σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή, ε, όποτε ξεκινά μια τέτοια συζήτηση, πολλώνεται. Και ε, αυτό διχάζει. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά το θέμα. Ε, Παρ' όλα αυτά πρέπει να συζητηθεί, διότι κοιτάξτε τι γίνεται στην Ευρώπη. 130 πυρηνικοί αντιδραστήρε. Και κάποια κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει να κλείσουν αντιδραστήρε. Ενώ άλλα κράτη-μέλη χτίζουν καινούριου. Ενώ μια τρίτη ομάδα διατηρεί όσου έχει. Γνωρίζω πόσο ακριβό και απαιτητικό τεχνολογικά ε, είναι να κλείσει ένας πυρηνικός αντιδραστήρας και θα πρέπει να γίνει επαρκής ε, έρευνα για την πυρηνική ασφάλεια έτσι ώστε αν διατηρήσουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες στην Ευρώπη αυτό να γίνεται με τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές. Και αυτό θα μας βοηθούσε να ε, εστιάσουμε με το σωστό τρόπο στο πρόβλημα και να ε, αποδραματοποιήσουμε την συζήτηση. Να την αποφορτίσουμε. Ε, γιατί ο κίνδυνος θα ήταν οι συζητήσεις αυτές να γίνουν εκτός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα ήταν λάθος, διότι εμείς έχουμε κανόνες για ασφάλεια, για την υγεία, έχουμε εμπειρογνωμοσύνη, τεχνογνωσία, έχουμε εμπειρογνώμονες ε, οπότε η, ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Πέρσι στην Πράγα ε, η συζήτηση έγινε και με την κοινωνία των πολιτών και με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις με μη κυβερνητικέ οργανώσει, με άλλου ενδιαφερόμενου και έτσι θα πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί η συζήτηση να περιοριστεί μόνο μεταξύ εμπειρογνωμόνων. Στην Πράγα η συζήτηση ήταν πολύ πιο πλατιά και κάλυψε πολλά ευαίσθητα ζητήματα. Η επόμενη ερώτηση αφορούσε την ε, προτυποποίηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Βρέθηκα στο Ανόμπερο πριν από δύο εβδομάδες περίπου. Δύο προϊόντα τράβηξαν την προσοχή μου. Πρώτον, μια επίδειξη ε, προς τον κύριο Μπάμα και την κυρία Μέρκελ που ήταν ένας φορτιστής που μπορούσε να φορτίσει την μπαταρία αυτοκινήτου για 500 χιλιόμετρα σε 25 λεπτά. Αυτό είναι εξαιρετικό επιτεύγμα. Είναι ήδη κατορθωτό σήμερα. Ο πρόεδρος είπε «Ελπίζω να έχετε το ίδιο πρότυπο και για τα αμερικάνικα αυτοκίνητα, για τις αμερικάνικες πρίζες. Του είπανε ναι εντάξει τα βόλτ ε, η τάση διαφέρει λιγάκι αλλά γενικά ναι. Δεύτερη επίδειξη σημαντική ήταν πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα ε, ως συσσωρευτές ενέργειας. Ε, στα ε, καινούργια κτίρια όταν θα έχουμε περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με ισχυρές μπαταρίες θα μπορούσαν αυτά τα, ε, ε αυτές οι μπαταρίες να ε, χρησιμοποιούνται για αποθήκευση ενέργειας η οποία αργότερα θα μπορούσε μάλιστα να πωλείται και στην, ε, ε, στην εταιρεία παροχής ενέργειας. Μα μου είπαν ότι οι μπαταρίες των αυτοκίνητων έχουν πέσει τα 1200 ευρώ, κάτι που μου φαίνεται εξαιρετική πρόοδος, θα εκτοξεύσει τις πωλήσει ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο μέλλον. Θα πρέπει οι ΗΠΑ και η Ευρώπη να υπογράψουν ένα μνημόνιο έτσι ώστε να καθοριστούν ε, δύο ε, εργαστήρια, Ίσπρα και Σικάγο, προκειμένου να συνεργαστούν για την ε, προτυποποίηση για την επεξεργασία προτύπων που θα αφορούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προκειμένου οι υποδομές να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη των πωλήσεων. Η επόμενη ερώτηση αφορούσε την επικύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει λόγους ε, να επιθυμεί αυτή η επικύρωση να γίνει το συντομότερο δυνατό. Θα προτείνω μια ανακοίνωση, θα υποβάλουμε μια ανακοίνωση για την μείωση του, α, της ε, χρήση ε, της, ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στα αυτοκίνητα και ταυτόχρονα θα ζητήσουμε ε, να επικυρωθεί σύντομο, το το δυνατό η Συμφωνία των Παρισίων. Ο κ. Γκερμπράντι ε, αναφέρθηκε στη συμπεριφορά των κρατών μελών που ε, ε αν, αντιδρούν μόνο με, τμηματικά. Η βιοενέργεια όμως είναι σημαντική ε, η Κομισιόν εκδίδει σύσταση, δεσμευτική σύσταση για τη βιομάζα και είναι ο τμήμα αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να βρούμε τρόπου έτσι ώστε η βιομάζα πράγματι να μειώσει τι εκπομπέ ε, αερίων θερμοκηπίου. Αυτό είναι ο στόχο μα και αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη βιομάζα, αυτή θα πρέπει να παράγεται με βιώσιμο τρόπο σε όλη την αλυσίδα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ε, επικαιροποιημένους λογιστικούς κανόνες, ε, κανόνες υπολογισμού μάλλον, να το πω έτσι, μέτρησης. Εργαζόμαστε επίσης για τα κριτήρια βιωσιμότητας της στερής βιομάζας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαβούλευση και για τα δύο αυτά ζητήματα. Ε, η συμμετοχή είναι πολύ ψηλή ήδη και την περσμένη εβδομάδα είχαμε μια πολύ επιτυχή συνάντηση μεταξύ των ενδιαφερομένων, των stakeholders. Τώρα εξετάζουμε τις αναλυτικές λύσεις για το πού θα μπουν τα κριτήρια. Η, το λογικό συμπέρασμα θα ήταν η, ε, η οδηγία ανανεώσιμων, αλλά θα μπορούσαν να μπουν και κάπου αλλού. Εξετάζουμε όλες τις αναλυτικές λύσεις. Να δούμε πού θα ενταχθούν αυτά τα κριτήρια. Σε ό,τι αφορά την καινούργια γενιά βιοκαυσίμων Σε αυτή τη φάση χρειαζόμαστε μια σταδιακή κατάργηση της πρώτης γενιάς βιοκαυσίμων. Ο λόγος είναι ο τρόπος με τον οποίο Πέδρασαν αρνητικά, η καλλιέργεια, στη γεωργία η καλλιέργεια των φυτών προορίζονταν για, τα, την πρώτη γενιά βιοκαυσίμων. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει τα πρώτη γενιά αυτή να καταρριφθεί σταδιακά. Αυτή τη στιγμή αναλύουμε το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μετάβαση προς πιο προηγμένα βιοκαύσιμα. Μία από τις ανακαινήσεις που προετοιμάζουμε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το διοξείδιο του άνθρακα ε, στι μεταφορέ, θα δίνει περισσότερε λεπτομέρειε για το πώ πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την περίοδο μετά το 2030, συμφωνώ κύριε Κερμπράντη με εσά. Θα πρέπει ήδη από τώρα να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε. Ο προγραμματισμό είναι σημαντικό, θα πρέπει η κοινή γνώμη να προετοιμαστεί, θα πρέπει να προετοιμάσουμε τι υποδομέ μα, τη βιομηχανία μα και βέβαια να προετοιμαστούμε για συμπεριφορικές αλλαγές στην κοινωνία μας. Αυτά βέβαια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και στα εθνικά σχέδια ενέργειας και περιβάλλοντος και κλίματος. Ε, για την δεκαετία 2020-2030 έχουμε καλά σχέδια, αλλά θα καλούμε τα κρατημέλη να κοιτάξουν και αυτά την περίοδο μετά το 2030. Διότι για να ε, τηρήσουμε τους στόχους του 2030 ήδη είναι δύσκολο το να προβούμε σε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις, 80-90% μέχρι τα μέσα του αιώνα, στα αέρια του θερμοκηπίου, θα είναι ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Οπότε θα πρέπει τα κράτη-μέλη ήδη να αρχίσουν να το σκέφτονται. Τι θα κάνουν μετά το 2030. Σε ό,τι αφορά τα επίσημα έγγραφα, γνωρίζετε πολύ καλά το επίσημο χρονοδιάγραμμα. Μέχρι το 2018 περιμένουμε το πάνελ του IPCC ε, να μας δώσει, να μας συμβουλεύσει πώς να ε, πετύχουμε το, το 1,5 βαθμό και μέχρι το 2030 έχουμε τις υποχρεώσεις μας από την όλη διαδικασία να προετοιμάσουμε ε, τον οδικό χάρτη για το 2050 και μέχρι το 2023 θα πρέπει να δούμε, να κάνουμε ένα απολογισμό πώς ε, σεβόμαστε και σε ποιο βαθμό σεβόμαστε τους ε, δείκτες και τις υποχρεώσεις μας. Ε, εκεί η Κομισιόν έχει να παίξει σοβαρό ρόλο, σας το υπόσχομαι. Η κυρία Κονέτσινα αναφέρθηκε σε τους στόχους που μερικές φορές αντιφάσκουν μεταξύ τους, δεδομένου ότι έχουμε διάφορες προκλήσεις το σημαντικό είναι να είμαστε λογικοί, ορθολογικοί και γι' αυτό πρέπει να σεβαστούμε την ιεραρχία των αποβλήτων. Πρώτον, να αποφύγουμε την δημιουργία αποβλήτων. Δεύτερον, να τα επαναχρησιμοποιούμε. Τρίτον, να τα ανακυκλώνουμε. Τέταρτον, αν όλες οι προηγούμενες εναλλακτικές λύσεις δεν υφίστανται να ε, χρησιμοποιούμε, να τα, να τα καίμε και να τα μετατρέπουμε σε ενέργεια. Και ασφαλώς ε, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύγουμε τους χώρους υγειονομικής ταφής, ε, την ταφή των ε, αποβλήτων μας γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τεχνολογίες αναπτυγμένες και για την ανακύκλωση και για την επαναχρησιμοποίηση και για την ε, καύση με παραγωγή ενέργειας. Η ταφή θα πρέπει να αποφεύγεται με κάθε κόστος. Ε, θα, η πρότασή μας ε, για την μετατροπή των αποβλήτων σε ενέργεια θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του χρόνου και θα λάβουμε υπόψη όλα τα προηγούμενα ανακοινωθέντα τα οποία έχουμε εκδώσει για την κυκλική οικονομία. Ελπίζω ότι θα βρείτε τις προτάσεις μας ισορροπημένες. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ. Περνάμε στο δεύτερο γύρο, η κυρία Γκροστέτα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε να μας ε, παρουσιάσετε την άποψή σας για αυτή την Ένωση για την Ενέργεια, ε, για την ενεργειακή απόδοση ε, και αποτελεσματικότητα, κάποτε, πάντοτε έχουμε την εντύπωση ότι δυσκολευόμαστε να τα ρυθμίσουμε όλα και όλα βέβαια εξαρτώνται και από τις επενδύσεις που γίνονται, που θα γίνουν. Μιλήσατε για την αεροπλοεία. Στον τομέα της αεροπλοείας υπάρχουν ήδη εταιρείε που καταβάλουν προσπάθειες και χρησιμοποιούν συγκεκριμένα είδη αεροσκαφών για συγκεκριμένα είδη διαδρομών, γιατί ήδη είναι πολύ πιο οικονομικά όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας σε αυτά τα αεροσκάφη. Γίνονται πράγματα. Το θέμα είναι όμως ε, τι θα επιβληθεί σε διεθνές επίπεδο. Γιατί δεν ε, θέλουμε πάλι να βάλουμε αυτό γκολ όπως κάνουμε τακτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα πυρηνική ενέργεια. Ευτυχώ που έχουμε την πυρηνική ενέργεια για να καταπολεμήσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ. Γιατί εδώ γνωρίζουμε ότι όσοι θέλησαν να σταματήσουν την πυρηνική ενέργεια, η μόνη είναι οι σταθμοί που λειτουργούν με άνθρακα. Ε, και μη χειρότερα ε, όσον αφορά τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα και την ποιότητα του αέρα. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχυθούν οι κανόνες ασφάλειας για την πυρηνική ενέργεια, αλλά την επόμενη δεκαετία δεν μπορούμε να μην το χρησιμοποιήσουμε για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τις αλλαγές, τις κλιματικές. Οι ανανεώσιμες ενέργειες, ωραία, τέλεια, αλλά δεν αρκούν για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Πρέπει να έχουμε και ένα κομμάτι πυρηνικής ενέργειας. Είναι απαραίτητο. Αλλά δεν μιλήσαμε για φυσικό αέριο, γιατί εγώ θέλω να σας μιλήσω γι' αυτό, γιατί στην Ένωση για την Ενέργεια υπάρχει και το φυσικό αέριο και η εξασφάλιση του ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Μιλήσατε για τη δημιουργία μιας ομάδας κατών μελών για να αντιμετωπίσουμε τις περιφερειακές ανάγκες. Ωραιότατα, αλλά πρέπει να έχουμε και μια ευελιξία. Διότι δεν πρέπει να περιορίσουμε το κάθε κράτος μέλος σε μια οργάνωση περιφερειακής συνεργασία μόνο, γιατί ε, θα ήταν πιο σκόπιμο να φτιαχτούν διάφορε διάφορες ομάδες περιφερειακής συνεργασίας με βάση τους ε, μεγάλους διεθνείς κινδύνους, ώστε ένα κράτος μέλος να μπορεί δηλαδή να είναι τμήμα πολλών περιφερειακών ομάδων. Και από ό,τι κατάλαβα θέλετε να αντικαταστήσετε τα εθνικά σχέδια διαχείρισης κρίσης από τα περιφερειακά. Πρόκειται για αντικατάσταση ή για καλύτερο συντονισμό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, Λάινεν. Ναι, κύριε Πρόεδρε. το τρίγωνο που μας παρουσιάσετε είναι καλό, εάν βγάλουμε και τα σωστά συμπεράσματα από τις προτάσεις αυτές. Τώρα συζητήσαμε πολύ για τις μεταφορές, όντως αυξάνονται οι εκπομπές στις μεταφορές, αλλά υπάρχει και μια άλλη συνιστόσα που είναι τα κτίρια. 75% της ορυκτής ενέργειας χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψήξη. Άρα χρειαζόμαστε και μια στρατηγική για heating και cooling. Οπότε ε, σήμερα στα νεόδημη τα κτίρια αυτό είναι πολύ πιο εύκολο ε, από αυτό που προέβλεπε η παλιά ε, οδηγία. Και εδώ και πέντε χρόνια συμμετέχω σε μια επιτροπή στην Ελβετία για την απονομή ενός βραβείου που έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα με το ίντερνετ, με ε, τις ε, τεχνολογίες επικοινωνίας και εμείς δεν επιτρέπεται να χάσουμε το τρένο. Μετά, τι γίνεται με χρηματοδότηση γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ενεχόμενοι εκεί στα κτίρια, υπάρχουν ιδιοκτήτες των κτίριων. Εκεί δεν είναι αρκεί το έψη το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, για την πράσινη χρηματοδότηση. Ασχολείται με πολύ μεγάλα έργα μόνο το έψη, όχι με αυτά τα μικρά. Τρίτο, η τεχνολογική επικοινωνία. Μόλις επιστρέφω από την Κίνα, έχουμε πάει με την αντιπροσωπεία εκεί και συζητήσαμε και για την πράσινη ανάπτυξη, φωτοβολταϊκά Κίνα, μπαταρίες Κίνα. Πού είναι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς πού θέλουμε να είμαστε ηγέτες και πώς μπορούμε να είμαστε και οι καλύτεροι ενδεχομένω ε, ή αν μη τι άλλο να παρακολουθούμε τις εξέλιξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Εγώ θέλω μόνο να υπογραμμίσω πόσο εκτιμούμε το γεγονός ότι έρχεστε εδώ και μας δίνετε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα υπόθηκαν για την Ενεργειακή Ένωση και εδώ και στην ανακοίνωση, στο ανακοινωθέν σας για την κατάσταση της ε, Ένωσης της Ενεργειακής για το 2015 και υπ' αυτό το φως θέλω να σας ερωτήσω τα εξής. Ένας από τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης είναι να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στα κρατημέλη και τα κρατημέλη της Ενεργειακής Κοινότητας όπως η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Βοσνία, η Ζωγαβίνη, η Σερβία, το Μαυροβούνιο κτλ. ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής ε, ε, Πολιτικής. Ποια είναι τα βήματα στα οποία προβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσει όντως αυτή τη συνεργασία. Και δεύτερη ερώτηση. Πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλουμε να έχουμε μια ένωση ότι, όπου τα κράτη-μέλη βλέπουν ότι αλεξαρτώνται για να έχουν ε, από ασφαλή ενέργεια προς τους πολίτες τους που θα βασίζεται σε πραγματική αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη. Αυτή ήταν μια παράθεση όπως ε, υπάρχει στο ανακοινωθέν σας για τη στρατηγική. Όμως, επικρατεί κάποιο διαρθωτικός διχασμός, δηλαδή έλλειψη εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, για την Ενεργειακή Ένωση. Για παράδειγμα, ανεπαρκείς δυνατότητες διασύνδεσης που δεν είναι πάντοτε τυχαία, κάποιες φορές είναι ηθελημένη, είναι σκόπεμη. Και επιπλέον, τα νέα κράτη-μέλη που εξαρτώνται υπερβολικά από το φυσικό αέριο της Ρωσίας είτε θέλουν να ανταγωνιστούν το βασικό του προμηθευτή, είτε θέλουν να διακινδυνεύσουν τις, είτε δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν τις συμφωνίες που έχουν κάνει ε, ατομικά, μεμονωμένα ο καθένας, εις βάρος της Ενεργειακής Ένωσης και μιλάω για το Nord Stream 2. Πώς θα δημιουργηθεί αυτή η τόσο απαραίτητη εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κρατη Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε, που ήρθατε για να συζητήσετε την άποψή σας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Κρότε μου πήρε την ερώτηση. Ε, ήθελα και εγώ να ρωτήσω ε, για αυτά που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μήνυ ε, πυρηνικούς αντιδραστήρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γι' αυτό τώρα θα κάνω άλλη ερώτηση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Ε, σας ερωτώ όμως, θα συμμετέχει και η Γεωργία, ιδιαίτερα με τη μείωση των πάρα πολύ μεγάλων ε, εκτροφών μονάδων εκτροφής, ε, στην κτηνοτροφία δηλαδή, που ε, εκπέμπει ε, πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα και γενικά ρηπαίνει. για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες θα ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι στόχοι των τρομοκρατών. Δεν θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Υπάρχει ένα ρίσκο τη στιγμή που συζητάτε για τέτοιου είδου πυρηνικά εργοστάσια. Ευχαριστώ, κύριος Μπελέτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλησπέρα σας. Πολλά ήδη υπόθηκαν για το ETS και τις τεράστιες προσπάθειες που έχουμε να καταβάλουμε και στην ε, μεταρρύθμιση. Και ο Πέτερ και ο Ματίας και ο Γκερμπλάντι ε, αναφέρθηκαν στην ε, ε, αεροπλοή. Τι θα γίνει με την κατανομή των προσπαθειών και τον καταμερισμό και στις μεταφορές, όχι μόνο στη οικοδομή, στα κτίρια. Θέλω να αφαιρθώ και στα βαρέα φορτηγά οχήματα και ε, στα λεωφορεία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία ε, και στι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ε, ε ενώ εμεί δεν έχουμε που θέλουμε να είμαστε και πρωτοπόροι. Δεν είναι δική μας φιλοδοξία λοιπόν να καταναλώσουμε πάρα πολύ χρόνο θα πρέπει πριν το 2030 να έχουμε αποτελέσματα και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Και για τη βιομάζα, εδώ στο Βέλιο που είναι και η πατρίδα μου, γίνεται μεγάλος λόγος για τη χρήση ε, τέτοιων εγκαταστάσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν στραγγαλιστεί, έχουν πεθάνει κυριολεκτικά τέτοια σχέδια πρόσφατα, γιατί γίνεται λόγος για την αποδοτικότητα, για τη βιωσιμότητα. Εμεί τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα για να επενδύσουμε στη βιομάζα, να εισάγουμε ξύλο, να εισάγουμε άλλα προϊόντα ή θα, θα επενδύουμε ε, στις ε, offshore ανεμογεννήτριε που είναι και πάρα πολύ ισχυρά επιδοτούμενες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ευχαριστώ κύριος ε, Παχνιό. Μάλιστα, κύριε την Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στην επικύρωση της συμφωνίας του στην κύρωση μάλλον τη συμφωνία του Παρισιού από τι ε, χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν δεσμεύτηκε να υποβάλει πριν από το καλοκαίρι δύο προτάσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η μία για την κύρωση τη συμφωνία των Παρισίων και η δεύτερη για την κατανομή των εθνική προσπάθεια ε, που θα έπρεπε να καναβάλει κάθε χώρα για να επιτύχει του ε, κοινοτικού στόχου για το πακέτο κλίμα 2030. Στι 3 Μαου η μάλλον η Νομική Υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μια, ένα σημείωμα για να αποσυνδέσει αυτά τα δύο θέματα. Διότι σήμερα αυτή η αποσύνδεση, μάλλον, ή μάλλον η σύνδεση μεταξύ των θεμάτων είναι προβληματική. Έχουμε την εντύπωση ότι τα κράτη-μέλη που εξαρτώνται από την καύσιμη ενέργεια, από την ορυκτή ενέργεια, δηλαδή Σλοβακία, Τσεχία, Πολωνία, ορίζουν την κύρωση της συμφωνίας αυτής από την ε, κατανομή των εθνικών προσπαθειών για να μειώσουν κατά τουλάχιστον 40% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030. Έχω την εντύπωση ότι η διαδικασία κύρωσης αυτής της συμφωνίας των Παρισίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία κρατείται όμοιρος από αυτές τις χώρες που εξαρτώνται από την ε, ρηκτή ενέργεια. Κύριε Αντιπρόεδρε, πώς μπορούμε να βγούμε λοιπόν από αυτήν την ομοιρία, τι θα κάνετε και πώς ε, θα μπορέσουμε να ε, κατανείμουμε έτσι την προσπάθεια, ειδικά σε μια φάση όπου βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις, να μπορέσουμε έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, πανέλθει, να σταθεί και πάλι στο ύψος των περιστάσεων και να μιλήσει με μια φωνή. Uh, ευχαριστώ πολύ. Πέτερλε. Ε, σας ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την πολλά υποσχόμενη εισήγηση με τις πολύ σαφές, σαφείς ιδέες. Το βιώσιμο μέλλον ε, απαιτεί μια συνεπή προσέγγιση σε διάφορα μέτωπα ταυτόχρονα. Με βάση τα όσα είπατε σε σχέση με τις πολιτικές εντός της Ένωσης, ε, θα ήθελα να τονίσω μια άλλη σημαντική πτυχή ή ευκαιρία που θεωρώ ότι είναι απαραίτητη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη, στρατηγική, τη συμφωνία στρατηγική ε, εταιρική σχέση και συμφωνίε με άλλου εταίρου στον κόσμο, ώστε να συμμετέχουμε στο πρασίνισμα των αναπτυσσόμενων του οικονομιών. Εγώ είμαι ικανοποιημένο από τι προθέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ αυτό τον τομέα όσον αφορά την Ινδία, αλλά υπάρχουν και άλλοι εταίροι. Όσο περισσότερο πρασινίζουμε τι εταιρικέ μα σχέσει, τόσο πιο κοντά θα φτάνουμε και στου στόχου των Παρισίων. Μπορούμε λοιπόν να μοιραστούμε τεχνολογία, εμπειρία, ε, εμπειρογνωμοσύνη. Μπορούμε, θα έλεγα, να μοιραστούμε και τις τρεις γωνίες του, ολόκληρο το τρίγωνο που αναφέρατε. Και οι ευρωπαϊκές τράπεζες αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόβλημα από λεφτά. Είναι η κατάλληλη στιγμή να τα χρησιμοποιήσουμε για, τους καλούς, για το σωστό σκοπό. Μπορείτε να επηρεάσετε τις εξελίξεις προς περισσότερες διατομιακές και πιο ολοκληρωμένες προσεκίσεις. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καμπεθόν Ρουίθ. Ασφαλώς και θα μιλήσω για την Ενεργειακή Ένωση, αλλά θα ήθελα να σχολιάσω πιο πολύ το όραμα. Γιατί ο στόχο είναι η προμήθεια, προμήθεια με ενέργεια στου καταναλωτέ και τη βιομηχανία. Ε, όλα αυτά ε, αναλύονται το πώς μπορεί να γίνει κυρίως και έχει γίνει λόγος και για την ενεργειακή απόδοση. Προφανώς γι' αυτό χρειάζεται συγκεκριμένη δέσμευση ο πλευράς των εθνικών κυβερνήσεων μέσω των εθνικών σχεδίων. Πρέπει όμως να αναλύσουμε και το κόστος ο πλευράς ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η, αρμοδιότητα βαρύνει κυρίως τα κράτη-μέλη αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλύει την κατάσταση. Δεδομένου ότι πάνω το 50% του, της τιμής της ενέργειας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φόροι και εισφορές. Ε, και δεν μιλώ μόνο για το κόστος της διανομής, αλλά γενικότερα τη φορολογική πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει μια συζήτηση για την δίκαιη φορολογική ενέργειας, έτσι ώστε πράγματι να είναι δίκαιη και βιώσιμη κοινωνικά. Επίσης θα πρέπει να εκδημοκρατιστεί ο εφοδιασμός, ο ενεργειακός εφοδιασμός και να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση αυτοκατανάλωσης, κατανάλωση δηλαδή της ενέργειας που παράγουμε εμείς ήδη. Τελευταίο σχόλιο, η ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας στην, στο Βέλγιο. Έχουμε ακούσει ειδήσει ε, τελευταία ε, για την ε, ε διανομή φαρμάκων με ιόδιο στον πληθυσμό προληπτικά και προφανώς υφίσταται κάποιος κίνδυνος, κάποια ανησυχία τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών. Ε, διαβάζοντας τον τύπο στη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, αυτό βλέπουμε. Ε, ορισμένοι πυρηνικοί αντιδραστήρες ε, που βρίσκονται σε κακή κατάσταση πήραν ε, αναβολή στο κλεισμό τους για 10 χρόνια, παρόλο που ήταν να κλείσουν το τέλος του χρόνου. Θα ήθελα να με ενημερώσετε για το ποιο είναι το επίπεδο ασφάλειας. Ευχαριστώ κύριο Μπάλτσο. Κύριε Επιτροπέ, δεν πρόκειται για άμεση ερώτηση, αλλά περισσότερο για έναν προβληματισμό. Όποτε έρχεστε εδώ στην Επιτροπή μας, δεν συζητούμε ποτέ το πώς η ε, ε, οι αποφάσεις επηρεάζουν τις τιμές. Πάντοτε μιλούμε για την κλιματική αλλαγή. Προφανώς αυτό, και αυτό αποτελεί αρμοδιότητά μας, αλλά η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την πυρηνική ενέργεια. Ακούσαμε ότι η, ε, η Επιτροπή θεωρεί πως το ενεργειακό μείγμα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και βέβαια, αλλά η Κομισιόν μπορεί να έχει τη δική της θέση για το θέμα. Ε, για παράδειγμα, προωθείτε τις ανεμογεννήτριες και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παρέμβαση σε, σε εθνικές αρμοδιότητες. Αλλά, δεν, αλλά το κάνετε παρόλα αυτά. Γιατί να μην το κάνετε και ως σύσταση ε, με την πυρηνική ενέργεια ένας Αμερικάνος ε, επιστήμονας έγραψε μια ανοιχτή επιστολή πριν από κάποια χρόνια για τα ωφέλη της πυρηνικής ενέργειας. Ε, και ανέφερε ότι η πράσινη, η πράσινη ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ε, από μόνες τους να λύσουν το θέμα, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής έλεγε ότι η πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να είναι ασφαλής, αλλά θα πρέπει να, σίγουρα υποχρεωτικά, αναγκαστικά να αποτελέσει τμήμα του ενεργειακού μείγματος για να πετύχουμε τους στόχους της κλιματικής αλλαγής. Οπότε φιλο, πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι σε σχέση με τη χρήση της, ε, των ανεσίμων πηγών ενέργειας, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστικοί σε ό,τι αφορά την επιτυχία των στόχων για την κλιματική αλλαγή. Δεν είναι δυνατόν η κλιματική αλλαγή ε, να ε, θεωρείται ε, του μείγματος και ξεπερασμένη. Κύριε Πίρικ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, ωραία αυτό που μας λέτε, αλλά ε, η Ολλανδική Προεδρία τα ξέρει αυτά που λέτε. Για την Ενεργειακή Ένωση, αφού μιλάμε για την ενέργεια, για την κυκλική οικονομία. Εδώ μπροστά σας ακριβώς κάθομαι απέναντί σας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλές εταιρείε που θέλουν. Εγώ είμαι από το Τβέντε. Έχουμε πάει ε, και έχει πανεπιστήμια, ε, έχει πολίτες, εταιρείε που ενδιαφέρονται, ε, αλλά δεν ξέρουν πώς να απευθυνθούν σε αυτό. Παράδειγμα, σε 700.000 ε, σπίτια, κατοικίες, νοικοκυριά θέλουν να αλλάξουν, ε, να ανακαινήσουν τα κτίρια για να είναι ε, ουδέτερα ως προς την ενέργεια. Πώς θα αποτανθεί ο κόσμος συγκεκριμένα, πώς θα βρει τον δρόμο για να φτάσει σε αυτό το στόχο. Και να ρωτήσω κάτι για τη γεωργία. Μιλάμε για την ε, συμφωνία για το κλίμα, αλλά η γεωργία κατά την άποψή μου δεν συμμετέχει ε, αρκετά. Εσείς στις δικές υπηρεσίες κάτι προετοιμάζετε. Ε, δεν αναφέρετε άμεσα, αλλά έμεσα τον κλάδο και εδώ πρόκειται για ε, πολλές θέσεις εργασίας κτλ. Και μιλάτε και για επιβολή φόρου. Σε πού θα βάλετε φόρο στη σόγια. Ο κόσμος ανησυχεί ε, σε κάθε συνεδρίαση ε, ε, ε, επαναλαμβάνω το ίδιο θέμα. Σε κάθε συνεδρίαση μιλάμε για την ε, επεξεργασία της ε, κοπριάς, για την ανακύκλωση. Το έχουν βάλει στα απόβλητα. Τι δουλειά έχει αυτό. Δεν είναι θέμα σκουπίδια, είναι ανακύκλωση για παραγωγή ενέργειας. Εγώ το θέτω κάθε φορά υπόψη σας. Ακούμε διάφορα παράπονα για την Ευρώπη, αλλά το και πέρα δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχετε εσείς για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ, ο Επίτροπος. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε από πού άρχισε ο δεύτερος γύρος, τα ονόματα. Από την κυρία Γκροστέτ. Μια στιγμή να τη βρω. Κάπου το έχω σίγουρα, έχω κρατήσει σημείο. <laughs> Here it is. I'm sorry. Thank you very much. Ε, ζητώ συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ, το βρήκα. Η κυρία Κροστέτ φυσικά αναφέρθηκε στην εναέρια κυκλοφορία και ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ήδη ε, κάνουν ε, οικονομίες, χρησιμοποιούν ειδικό καύσιμο ε, και προσέχουν το περιβάλλον, ενώ άλλε αεροπορικέ εταιρείε αδιαφορούν. Οι Ευρωπαϊκέ είναι από τι καλύτερε τι επιδόσεις τους σίγουρα και δεν είναι τεράστια επιβάρυνση να συμμετέχει ε, σε μια τέτοια προσπάθεια και στο ευρωπαϊκό σύστημα και ο κλάδο τη ε, νέρης, κυκλοφορίας των αερομεταφορών. Όταν πρόκειται για ε, τα αέρια του θερμοκηπίου. Υπάρχει βελτίωση Αλλά τι γίνεται με τις υπόλοιπες εταιρείε ε, αερομετοφορών παγκόσμιες, διεθνείς που ε, πετάνε πάνω από την Ευρώπη και πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα. Για την ε, πρόταση αυτή σήμερα πρέπει να πω ότι αλλάζει η κατάσταση. Σιγά σιγά βελτιώνεται η κατάσταση αυτή μεταξύ των μεγαλύτερων εταιριών και όλες οι νέες εξελίξεις εντός του ΑΕΚΑΟ μας κάνουν να είμαστε πιο αισιόδοξοι και να ε, συνεργαστούμε για, ε, για θετική συμφωνία τον Οκτώβριο. έτσι ώστε μέχρι το 2020 να μειωθεί η συμμετοχή τους ε, στην εκπομπή διοξιδίου και γενικώ αερίων θερμοκηπίου. Προχωρούν και οι τεχνολογικές εξελίξεις και αυτό μας επιτρέπει να προχωρούμε ταχύτερα. Βασική ερώτηση όμως της κυρίας Γκροστέτ ήταν η περιφερειακή συνεργασία και η ενεργειακή ασφάλεια ε, στον εφοδιασμό. Να σας εξηγήσω γιατί το προτείνουμε αυτό. Είδαμε στο παρελθόν ότι ιδιαίτερα στον τομέα ε, του φυσικού αερίου διαπιστώσαμε ότι τα κράτη-μέλη όταν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα ε, μόνα τους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μιλώ για τα περισσότερα ε, κράτη ε, που είναι μικρά ή μεσαία στο μέγεθος. Πέρασαμε μια κρίση το 2006, μια άλλη το 2009, κάναμε αυτά τα stress test, τις δοκιμές αντοχής και τα κράτη που είναι τα πιο εκτεθειμένα, πώς θα αντιμετώπισαν το πρόβλημα, τους βοήθησαν οι γείτονες. Βάλαμε πέντε κριτήρια. Γεωγραφική εγκύτητα, σχέση, συστήματα διασύνδεσης, αποθήκευση φυσικού αερίου, ε, συνεργασία ε, των φορέων διαχείρισης και τέτοια κριτήρια για να μπορούν να συσταθούν αυτές οι γεωγραφικές ομάδες. Παρακολουθήσαμε πολύ στενά και τη συζήτηση που γίνεται μεταξύ των κρατών μέλων και είναι γεγονό ότι ιδιαίτερα τα μεγάλα κράτη-μέλη είναι πολύ μεγάλα για να συμμετέχουν σε μία και μόνο ομάδα. Αυτή την εντύπωση έχω αποκομίσει και αυτή την αίσθηση. Είναι προσωπική η παρατήρηση. Και αυτό που έχει σημασία και για μένα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να βεβαιωθούμε ότι όταν εγκρίναμε την οδηγία για την ασφάλεια του εφοδιασμού, θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι γείτονε ε, και οι περιφερειακοί εταίροι θα πρέπει να συνεργάζονται για να έχουν σχέδια αντιμετώπισης μιας επίγουσας κατάστασης σε μια ολόκληρη περιφέρεια. Ποια είναι τα προπετούμενα, πώς έχει η διασύνδεση, τι επίπεδα ε, αποθήκευση ενέργειας χρειαζόμαστε για να βοηθηθούν αυτές οι χώρες. Το ίδιο ισχύει και για τη Δυτική Ευρώπη και για την Νότια Ανατολική, όχι μόνο για την Ανατολική. Χρειαζόμαστε λοιπόν περιφερική συνεργασία. Ενδεχομένω τα μεγάλα κράτη μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες περιφέρειες. Αυτό δεν πειράζει νομίζω, απλώς να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχουν σχέδια αντιμετώπισης μιας επίγουσας κατάστασης για όλη την Ευρώπη, για να είναι καλά ανεπτυγμένα, ρεαλιστικά ε, φτιαγμένα και να λύνουν τα προβλήματα. Γνωρίζω ότι αυτή η συζήτηση τώρα είναι πάρα πολύ έντονη για το θέμα αυτό. Ελπίζω να βρούμε καλές λύσεις και για την πρόταση αυτή, διότι όπως γνωρίζετε, γνωρίζετε συγγνώμη, έχουμε συμπεριλάβει στο παράρτημα τις περιφερειακές ομάδες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι βασικός πυρήνας της πρότασης, δηλαδή να είναι υψηλή ποιότητας ε, η αντίδρασή μας ε, στις επίγουσες καταστάσεις. Δεν μπορώ να έψω την έκβαση. Είναι περίπλοκο. Αλλά εμείς να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα να μπορεί σε κάθε περιφέρεια, κάθε κράτος μέλος να τρέχει και να το βοηθούν οι γείτονες. Ε, η δεύτερη ερώτηση ήταν τον κύριο Λάινεν. για τη θέρμανση, τη ψήξη και τα κτίρια. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι αυτή μια από τις ε, πρώτες προτεραιότητες του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και την ε, κόστη και κατανάλωση της ενέργειας, γιατί είναι γνωστό ότι το μίμηση της κατανάλωσης ενέργειας αφορά την ψήξη και τη θέρμανση των κτηρίων. Θα μπορούσαμε να τα πάμε πολύ καλύτερα λοιπόν εκεί. Α, λοιπόν όχι μόνο αναθεώρηση της οδηγίας για την ε, απόδοση της ενέργειας, την επάρκεια μάλλον της ενέργειας, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και λίγο πιο πέρα, να δούμε πώς αυτά τα κτίρια όχι μόνο θα είναι ε, επαρκεία ενεργειακά, αλλά και ευφυή. Τα νέα και ανανεωμένα κτίρια να είναι κομβή, να, είναι, να συνδέονται μεταξύ τους μέσα σε αυτήν την ολοκληρωμένη υποδομή, ώστε να μπορούμε να ε, παράγουμε ακόμα και ενέργεια, αλλά και να συλλέγουμε ενέργεια μέσω των κτηρίων. Μια ευφυή υποδομή με διασυνδέσεις όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μπορούσαν να φορτίζονται ή ενδεχομένως να έχουμε και πύργους ε, αναμετάδοσης για τα ε, σήμα Wi-Fi. Θα πρέπει να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά, γιατί θα χρειαστούμε αν θέλουμε να έχουμε κινητικότητα άνευ στο μέλλον. Αυτό λοιπόν που κάνουμε και προσπαθούμε να ε, εντοπίσουμε σε αυτό, να εστιάσουμε σε αυτό στην Κομισιόν είναι να έχουμε αυτά τα benchmarks, ε, κάποιους στόχους που να εντοπίζονται όχι μόνο ως ε, επαρκής από άποψη ενέργεια, αλλά και ευφυής, γιατί είναι ένα νέο στοιχείο αυτό και εξετάζουμε το κατά πόσο θα μπορέσουμε να το συμπεριλάβουμε σε αυτή την πρόταση, να τη διευρύνουμε κάπως, γιατί αυτά ακούμε πολύ από τους δημάρχους, δηλαδή να δούμε πέρα από την επάρκεια της, ε, ε, της ενέργειας, να δούμε και πώς θα καταστήσουμε πιο ευφυείς τις υποδομές μας, τις πόλεις μας. Και φυσικά και ευφυή χρηματοδότηση και να δούμε πώς θα εξετάζουμε όλα τα προγράμματα που είχαμε στην Κομισιόν και που κατά κάποιο τρόπο συνδέονται με αυτή την ε, ατζέντα. Διαρθωτικά ταμεία ή μικρότερα προγράμματα που είχαμε στην DG Ενέργεια, στην DG Regio και όλα να τα βάλουμε στην ίδια, στην ίδια θηρίδα. Και μετά το ΕΦΣΙ, το πρόγραμμα επενδύσεων του Juncker, γιατί είδαμε πόσο επιτυχές ήταν. Ήδη επενδύθηκαν 100 δις σε λιγότερο από ένα χρόνο και να δείξουμε ότι αυτό ήδη είναι ένα σχήμα που μπορούμε να μοχλεύσουμε σημαντικούς πόρους ε, για την προσπάθεια εξυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να αντλήσουμε και από τα τους θεσμούς πράσινης χρηματοδότησης. Έχουμε ήδη επαφές με διάφορα ταμεία, ιδρύματα και αυτό που μου έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό είναι μια συνάντηση όπου οι συμμετέχοντες ε, ανέφεραν τα 9 τρισεκατομμύρια ευρώ που ελέγχουμε και θέλουν και να επενδύσουν και στο μέλλον σε πράσινα projects, σε πράσινα μακροχρόνια projects, μακροπρόθεσμα projects. Δεν είμαστε λέει τράπεζες, είμαστε επενδυτικά ταμεία. Χρειαζόμαστε κάποιον να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή και να μπορέσουμε έτσι να επενδύσουμε σε αυτά τα projects. Ε, να έτσι να δημιουργήσουμε λοιπόν ε, την ε, δυνατότητα για επάρκεια και χρήση της ενέργειας. Τώρα, νομίζω ότι ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι μπορέσαμε να φέρουμε στην ε, καθημερινή πολιτική το θέμα της πράσινης ενέργειας και των πράσινων πολιτικών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προσπαθούμε να δείξουμε, από όλε τις παγκόσμιες οικονομίες μπορούμε να δείξουμε, προσπαθούμε να δείξουμε στους άλλους ε, εταίρους μας ότι μπορούμε να αναπτυχθούμε και ταυτόχρονα να μειώσουμε τις εκπομπές. Ε, μόνο εμείς, μοναδικοί είμαστε, μόνο εμείς θα έχουμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό. Και στην πορεία έχουμε χτίσει ένα τεράστιο όγκο τεχνολογικό και ανάπτυξη ευρεσιτεχνίε, γνώση, εμπειρογνωμοσύνη για το πώ το καταφέρνουμε αυτό. Να εστιάσουμε λοιπόν την προσοχή στην τεχνολογία τη μπαταρία, στην ε, αιωλική ενέργεια, την αιωλική τεχνολογία κτλ. Πού θέλουμε να είμαστε πρώτοι λοιπόν στην Ευρώπη, να μπορέσουμε να κυριαρχήσουμε πιστεύω στην σορευμένη γνώση από αυτή την ενεργειακή μετάβαση. Πρόκειται για τεχνολογική τεχνογνωσία που έχουμε οικοδομήσει στη διάρκεια των ε, χρόνων για το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη νέα τεχνολογία. Και αυτό είναι πολύ ε, απαιτητικό. Υπάρχει ζήτηση στην αγορά για το πώς θα γίνουν τα συστήματα πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά για χρήση όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά για ολόκληρη την ε, κοινότητα, την παγκόσμια κοινότητα. Σελίμοβιτς, ρωτήσατε για τη συνεργασία με την ε, κοινότητα της ενέργειας. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι η Ενεργειακή Ένωση δεν σταματά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ακριβώς εννοούσαμε ότι θέλαμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία και στις χώρες της ενεργειακής κοινότητας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε από νομικής άποψης πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε την ενέργεια σε ένα σωστό νομικό πλαίσιο και νομίζω πως η Γραμματεία της Επιτροπής Ενέργειας κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε πως χώρες όπως η Ουκρανία υιοθετούν νέο μοντέλο νέους κανόνες και νέα σύγχρονη νομοθεσία που την εντάσσουν στα συστήματά τους. Είναι η προτεραιότητα αυτή για το μέλλον. Δεύτερη σημαντική προτεραιότητα είναι να εξετάσουμε αυτή την γειτονία, μάλλον να τη θεωρήσουμε ως έναν ευρωπαϊκό χώρο συνεργασίας να φτιάξουμε δηλαδή διασυνδέσεις, interconnectors, να είμαστε κοντά όχι μόνο στα PCIs αλλά και στα projects που ονομάζονται PESIs, δηλαδή projects κοινού συμφέροντος για την ενεργειακή κοινότητα πώς προχωρούμε εκεί και μετά να δουλέψουμε και πάνω στις προκλήσεις που παρουσιάζονται από δύο χρηματοδοτικά μέσα. Από τη μία έχουμε την ευρωπαϊκή πλευρά και από την άλλη έχουμε το μέσο για τη γειτονία. Είναι όμως κάτι το εφικτό. Ε, πρέπει να δούμε απλά πώς θα προχωρήσουμε. Όσον αφορά τώρα την έλλειψη εμπιστοσύνη στην Ενεργειακή Ένωση και το ρυθμό οικοδόμησης των, των διασυνδέσεων, interconnectors, Είδατε ότι 11 χρόνια πήρε να φτιάξουμε ένα, μια, ένα στην Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι είτε τεχνικά είτε οικονομικά. Πάντως έχετε δίκιο ότι κάποια ζητήματα ξεπερνούν αυτά τα εμπόδια και αφορούν περισσότερο την ανησυχία της, του ανοίγματο τη ε, χώρε αγοραστή, στην ανταγωνισμό του φυσικού αερίου ή στην ηλεκτρισμό που έρχεται από άλλο κρατό μέλο. και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε γιατί ε, πραγματικά θέλουμε, πρέπει να δουλέψουμε να υπάρχει ελεύθερη ροή ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εφόσον θέλουμε να υπάρχει ενεργειακή ένωση πρέπει να δουλέψουμε σε διάφορα επίπεδα ώστε οι interconnectors να κατασκευαστούν. Ε, και για το θέμα του Nord Stream αναφέρθηκα σε αυτό για το πόσο σημαντικό είναι να σεβόμαστε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για περί ενέργειας, περί περιβάλλοντος, περί δημοσίων κατοικών ε, διαγωνισμών <clears throat> ώστε να βρούμε μια λύση ώστε η διέλευση για την Ουκρανία να διατηρηθεί. Διαφορετικά θα ήμασταν ενάντια σε όλες τις προσπάθειες και πολιτικές που έχουμε προς αυτή τη χώρα που εξακολουθεί να περνά αναταράξεις και εντάσεις. Και βεβαίως πρέπει να αποφύγουμε την πόλωση που φέρνει αυτό το project στην Ένωση. Γι' αυτό και αναπτύσσουμε διάφορα project και στρατηγικές. Ελπίζουμε ότι θα βρούμε μια καλή ευρωπαϊκή λύση και σε αυτή την πρόσκληση. Τώρα, κλιματικές αλλαγές, γεωργικός τομέας και κτηνοτροφία. Πρέπει να βρούμε μια λογική λύση για το, κατα... για το πόσο γεωργικός τομέας θα μπορέσει να συνεισφέρει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ε, με έναν ε, εύλογο τρόπο. Γνωρίζουμε τους περιορισμούς, γνωρίζουμε τις τεχνικές ε, δυνατότητες και λύσεις, ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες των χωρών στις οποίες αυτή η τομή είναι ισχυρή, οπότε πρέπει να βρούμε μια ισορροπημένη πρόταση την οποία να μπορούμε να εφαρμόσουμε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τους μικρούς ε, σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Ε, δεν μίλησαμε για τον Ίτερ σήμερα που είναι ένας, ε, ένα έργο, τεράστιο έργο σύνδεξης. Στηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Οι, οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες αναφέρονται στην, στις προτάσεις για την πυρηνική έρευνα και από, το, το, από την Breakthrough Coalition του Bill Gates οικονομικά. Ε, υπάρχει μια ομάδα ε, ε, επιστημόνων που κάνουν τέτοιου είδους έρευνα στην Ευρώπη. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να σεβαστούμε τις εθνικές αποφάσεις περί του ενεργειακού μείγματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα φορτηγά και τον τομέα των μεταφορών, Έχετε δίκιο. Στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, τα φορτηγά ε, είναι όχι μόνο πιστοποιημένα, αλλά ε, ε, συμμορφώνονται και με συγκεκριμένα όρια. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μου. Θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό το 2017. Η ημερήσια διάταξη φέτος είναι ήδη αρκετά φορτωμένη. Ήδη σκεφτόμαστε να εισάγουμε την ε, διαδικασία παρακολούθησης και πιστοποίησης, πιστοποίησης και παρακολούθησης, να ξέρουμε τι κάνουν, τι επιδόσεις έχουν τα φορτηγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η απόδοσή τους ό,τι αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Πρέπει να διαθέτουμε αρκετά στοιχεία για να επεξεργαστούμε μια πολιτική απόφαση στο μέλλον. Τώρα, βιομάζες και ε, ε, offshore. Λοιπόν, για τη βιομάζα. Αν μιλούμε για βιομάζα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνες μας είναι επαρκείς. Οι κανόνες μέτρησης δηλαδή, έτσι, διότι δεν θα πρέπει για να πετύχουμε εμείς τους στόχους μας εδώ να καταστρέφουμε τα δάση αλλού. Με καλές ε, προθέσεις μπορούμε να δημιουργήσουμε περιβαλλοντικό χάος και περιβαλλοντική καταστροφή αλλού παρόλε ενώ τι καλέ μα προθέσει. Οπότε πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχονται, πού προέρχεται η βιομάζα και αν είναι πραγματική βιομάζα. Δεύτερον, διαχείριση των δασών. Η χρήση της βιομάζας θα πρέπει να γίνεται με βιομάζα που προέρχεται από βιώσιμα δάση που ε, την χάνουν επαγγελματικής διαχείρισης. Αυτό είναι ε, εκ των όνου κάνευ όρος προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η βιομάζα την οποία χρησιμοποιούμε εδώ αντιστοιχεί σε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Θα πρέπει να, χρησιμοποιηθούν, να χρησιμοποιούνται σύγχρονοι τρόποι διαχείρισης των δασών και των καλλιεργειών. Offshore. Ε, η υπεράκτεια ε, παραγωγή ενέργειας, ε, η παραγωγή στη θάλασσα. Σε δύο εβδομάδες θα, θα συναντηθούμε με τις χώρες που θέλουν ε, να αναπτύξουν ε, το δίκτυο της βόρειας θάλασσας στη θάλασσα, με παραγωγή ενέργειας στη θάλασσα. Είναι ένας τομέας ο οποίος έχει τρομακτικό δυναμικό, έχει πολλές δυνατότητες. Θα πρέπει οι λύσεις που θα επιλέξουμε να είναι αποτελεσματικές, αποδοτικές ό,τι αφορά τη σχέση κόστους-οφέλους. Θα πρέπει τα δίκτυα παραγωγής ενέργειας στην ανοιχτή θάλασσα να συνδέονται ε, με το κεντρικό δίκτυο της υπηρετικής ε, Ευρώπης ε, γιατί αλλιώς το κόστος κινδυνεύει να είναι πολύ ψηλό. Κύριε Παρνιού, αναφερθήκατε στο κατά πόσον ορισμένες χώρες που εξαρτώνται από την παραγωγή άνθρακα, παραγωγή ενέργειας από άνθρακα, θα θέσουν υπομοιρία την Συμφωνία των Παρισίων. Δεν το νομίζω. Άκουσα στη Νέα Υόρκη όλους τους ε, αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, που κατέστησαν σαφές πως χρειάζεται να επικυρωθεί η Συμφωνία των Παρισίων το συντομότερο δυνατό. Ορισμένες από αυτές τις χώρες προφανώς θέλουν να δουν πρώτα ποιε είναι οι συγκεκριμένε νομοθετικέ μα προτάσει. Γι' αυτό το λόγο βιαζόμαστε. Ήδη υποβάλαμε το ETS. Ε Τώρα έχουμε τη Συμφωνία του Παρισιού, έτσι ώστε να καταστήσει σαφέ τι προτείνουμε στα κράτη-μέλη και στον τομέα ο οποίος δεν καλύπτεται από το εμπόριο ε, ε, ε, ε το ETS το εμπόριο εκπομπών. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ε, υποβάλουμε τις προτάσεις μας για να ε, γνωρίζουν όλοι ποιο είναι το πανόρμα για τα επόμενα χρόνια. Πριν από μερικές εβδομάδες το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε η Συμφωνία του Παρισιού να επικυρωθεί από όλους το συντομότερο δυνατό. Και ε, προτείνατε την ε, πρασίνηση των στρατηγικών συμφωνίων όπως για παράδειγμα με την Ινδία. Σίγουρα αυτό θα γίνει στο μέλλον. Ε, θα, θα είναι ο κανόνας στο μέλλον. Οι εμπορικές ε, συμφωνίες είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στην Αφρική για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και θα πρέπει να μάθουμε και από την μόχλευση του, ταμείου, ε, του Ταμείου Juncker έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε κάτι παρόμοιο και στην Αφρική για να στηρίξουμε την, τον εξυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα και την πρασίνησή του. Μετά, εθνικά σχέδια και ευάλωτες ομάδες πολιτών, καθώς επίσης και το κόστος. Το φθινόπωρο φέτος θα ξεκινήσουμε συζητήσεις προκειμένου να υποβάλουμε μια έκθεση σε συνεργασία με το Eurostat για την ε, τιμολογιακή δομή της ενέργειας σε κάθε κράτος μέλος. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει Είναι, ε, και πρέπει να γίνει έντιμα για να δούμε τι ακριβώς συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ενέργειας. Ε, Ε, έχουμε σημαντικά πλεονάσματα και ταυτόχρονα πολύ υψηλέ ε, τιμές ε, στον τελικό καταναλωτή. Κάτι που δέχεται πολλές επικρίσεις. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος διανομής, διάφοροι φόροι και τέλη, ένα κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής των κρατών. Θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε την τιμολογιακή διάρθρωση τις ενέργειες σε κάθε χώρα, να δούμε πώς αυτή μπορεί να γίνει πιο δίκαιη και πιο διάφανη κυρίως, πιο διαφανής, προκειμένου επίσης ε, να εξασφαλίσουμε τον εκδημοκρατισμό της παραγωγής ενέργειας και να δώσουμε περισσότερη εξουσία στους πολίτες αν θέλουν να χρησιμοποιούν περισσότερη λιγότερη ενέργεια. Η κατάσταση στο Βέλγιο. Παρακολουθούμε πολύ κοντά, από πολύ κοντά την ε, ε, κατάσταση. Γνωρίζουμε τις ανησυχίες των γειτόνων. Είμαστε σε επαφή με τις βελικές αρχές, διότι η φυσική και λειτουργική ασφάλεια είναι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μεγάλο βαθμό, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε σε επαφή με τις βελικές αρχές, τις ενθαρρύνουμε να συζητούν τα ζητήματα αυτά και με τους γείτονες έτσι ώστε και οι γείτονες χώρες να γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση ασφάλειας στο Βέλγιο και ε, να ε, μην ανησυχούν. Ένα παρόμοιο ερώτημα αφορούσε την τιμολόγηση και τη σημασία της τιμολόγησης. Είναι αλήθεια ότι για τη βιομηχανία και για τους πολίτες ένα ε, Κάτι που πολύ συχνά συζητείται είναι η τιμή της ενέργειας και πώς αυτή συγκρίνεται με άλλους ανταγωνιστές ή με άλλες χώρες. Στην έκθεση στην οποία αναφέρθηκα, ε, απαντώ στην κυρία Καπεθόν Ρούιθ, ε, θα αναφερθούμε σε αυτά τα θέματα. Σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια, νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό που έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται σε πολλά κράτη-μέλη. Να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ενέργειας όλο, όλο, να συμπεριλαμβάνονται όλα τα κόστη. Το κόστος κτισίματος κατασκευής των πυρηνικών σταθμών, το κόστος παραγωγής ενέργειας και το κόστος εγκατάλειψης κλεισίματος ε, των πυρηνικών σταθμών. Μόνο έτσι θα ξέρουμε πώς συγκρίνεται το κόστος πυρηνικής ενέργειας με το κόστος των άλλων τύπων ενέργειας. Η τελευταία ερώτηση αφορούσε την κυκλική οικονομία και την γεωργία και εκτενοτροφία καθώς επίσης και τα απόβλητα αυτού του τομέα. Η κυκλική οικονομία, για την κυκλική οικονομία είχαμε αναφερθεί στην ανακοίνωσή μας σε διάφορες αρχές και εναλλακτικές λύσεις, τις οποίες θα λάβουμε υπόψη όταν κάνουμε τις τελικές μας προτάσεις πριν το τέλος του χρόνου, όπως έχουμε υποσχεθεί. Ο τομέας της γεωργίας ε, θα είναι ένα βασικό κομμάτι των προσπαθειών μας ε, ε, που θα συγκεκριμενοποιηθούν μέσω της πρότασής μας για τον διαμοιρασμό της προσπάθειας. Θα πρέπει να δούμε πώς, τι βάρος θα αναλάβει κάθε τομέας, κάθε κλάδος. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα τόσο πολύ να απαντήσω, αλλά ήταν πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε για την παρουσία σας σήμερα εδώ ενώπιον μας, για το διαρθωμένο διάλογο, αλλά και για τις λεπτομερείς εμπεριστατωμένες απαντήσεις που δώσατε. Σας ευχαριστώ. Ε, θα τα ξαναπούμε. Πάμε αμέσως στο επόμενο θέμα στη Μέση Διάταξη, γιατί έχουμε καθυστερήσει προτείνω να περάσουμε μέσω στα σημεία 6 και 7, σημεία στις διάθεση, στο καλό να πάτε, ε, που είναι ο προπολογισμός του 2017 και η εντολή για το τριμερή διάλογο, καθώς επίσης και ανταλλαγή απόψεων με το Γιάννη Γκάιερ, Γενικό Εισηγητή για το Σχέδιο Προπολογισμού 2017. Φέτος ξέρετε ότι έχει αλλάξει κάπως η διαδικασία και μάλιστα πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα έτη για τον εξή απλό λόγο. Τώρα είμαστε στο σχέδιο προπολογισμού, ε, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να περιμένει το δημοψήφισμα για το Brexit πριν ε, δημοσιοποιήσει ε, το σχέδιο προπολογισμού. Θα δώσω όμως αμέσως το λόγο στο Γενικό μας Συγητή για να μας εξηγήσει τη θέση του για το προπολογισμό του 17 και μετά θα αρχίσει η συζήτηση για το βασικό θέμα στη μέση διάταξη που είναι πιο σημαντικό για την Επιτροπή ΕΜΒΗ του 2017. Ο κύριος Γκάιερ έχει το λόγο. Και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά να είναι Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πάντα μεγάλη ευχαρίστηση για μένα να ακούω το Μάρο Σεφσκοβίτς, οπότε πραγματικά απίλαυσα αυτή τη συζήτηση. Ε, να δεχτώ την πρόσκλησή σας να σας ε, παρουσιάσω συντομία ε, τη ε, σκέψη μου για τον προπολογισμό. Στην Ολομέλεια του Απριλίου στο Στρασβουργό, με μεγάλη πλειοψηφία, ε, ε, εγκρίναμε τις κατευθυντήριες γραμμές, τις οδηγίες για τον υπολογισμό του 2017 αν μου επιτρέπετε να σας τις παρουσιάσω σε σημαντικότερα σημεία επιγραμματικά εν είδη τίτλων. Γιατί οι διαπραγματεύσει για το προϋπολογισμό θα γίνουν έτσι πιο διαρθρωμένες με βάση αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές. Ε, πρώτον, θέλω να πιστήσω την προσοχή σας ότι στις διαπραγματεύσεις του προπολογισμού για το τρέχον έτος, το 2016, τα περιθώρια που είχαμε, ιδιαίτερα στην κατηγορία 3, που αφορούν μέρη και τα προγράμματα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, τα εξαντλήσαμε 100%. 100%. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Στο τίτλο και την κατηγορία 3 έχουμε πάρα πολλά μέτρα εσωτερικής πολιτικής που πρέπει να χρηματοδοτούνται από εκεί και που δίνουν ε, χρήματα στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την προσφυγική κρίση. Έχουμε τώρα μια κατάσταση που έχει ως εξής. Αφενός όλες οι κρίσεις που αφορούν το προπολογισμό του τρέχοντος έτους συνεχίζονται και του χρόνου. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα αλλάξει η κατάσταση στο προσφυγικό, ε, δηλαδή ότι του χρόνου θα χρειαστούμε λιγότερα χρήματα επειδή θα αποκλιμακωθεί. Θα συνεχιστεί και η οικονομική κρίση που σοβεί σε διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου ε, με ένα μεσοπρόθεσμο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε. Ένα τέτοιο πλαίσιο για το οποίο πολλά κράτη-μέλη χάρηκαν και η χώρα από την οποία κατάγομαι εγώ, το λέω ηρωνικά τώρα, μεγάλη πολιτική επιτυχία που ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά περιορίζεται, περικόπτεται αντί να αυξάνεται. Και τώρα, και δεν το λέω ηρωνικά, ε, αυτά που λέγαμε για τα χρήματα από ε, το 2013 ήταν ωραία λόγια, αλλά σήμερα δεν είμαστε σε θέση να δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά χρήματα για να αντιμετωπίζει τις κρίσεις που μας βρίσκουν σε κάποιο βαθμό. Ήδη έχουμε συμπληρωματικό προϋπολογισμό από τούτη την εποχή τώρα που δεν έχει προχωρήσει το έτος, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολιτικές προκλήσεις να αντιμετωπίσει και δεν φτάνουν τα χρήματα. Δηλαδή από το μήνα Μάιο ήδη έχουμε διορθωτικό και συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Το πολιτισμο δημοσιονομικό πλαίσιο μας δένει τα χέρια και ε, στην κατηγορία 3 και ειλικρινά δεν είμαι καθόλου βέβαιος τι θα γίνει μέσω πρόθεσμα και αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε την προγραμματική περίοδο. Γι' αυτό στα τέλη του έτους επίκειται, όπως ξέρετε, μια αναθεώρηση μετά από πρόταση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την περιμένω αυτή με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. 3,38 δις επίσης πρέπει να βρούμε για εγγυήσεις για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Δεν έχουν ακόμα κινητοποιηθεί τα κονδύλια αυτά επαρκώς όλα. Οπότε βλέπετε πως έχει κατάσταση και ήρθε εδώ η πρόταση από τις κατευθυντήριες γραμμές να συνδέσουμε ε, τις οικονομικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα μέσα του προϋπολογισμού για να βρούμε ε, προστιθέμενη αξία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό τουλάχιστον στην οικονομική πολιτική. Έχουμε και άλλα ε, βαριά προγράμματα που θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε, η πρωτοβουλία για την απασχόληση της νεολαίας, η καταπολέμηση της φτώχειας και η προστασία του κλίματος. Είναι πολλά αυτά που καλείται να καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν φτάνουν τα λεφτά, γιατί έχουμε λιγότερα χρήματα από ό,τι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αυτά είναι τα πλαίσια πάρα πολύ σφιχτά. Ο κύριος Λαβία είπε προηγουμένως, και τώρα το ξαναλέω ηρωνικά, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστερεί να καταθέσει το σχέδιο υπολογισμού λόγω του Βρετανικού δημοψηφίσματος. Αυτό ε, το διαψεύδει μαζικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατηγορηματικά, γιατί η επίσημη θέση είναι ότι εντάξει υπολογίζουμε τώρα ε, τα χρήματα που χρειάζονται για το προσφυγικό. Κάτι τέτοια λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως δικαιολογία. Αλλά φυσικά ο λόγος είναι αυτός που είπατε, ο κρίσιμος και ο αποφασιστικός. Και εμένα δεν με ικανοποιεί αυτή η δικαιολογία. Στον Περλεμό, ε, αυτή τη στιγμή στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε καν τις πόρτες δεν χτυπάνε, μην τυχόν και τρομάξει κανένας βετανός ψηφοφόρος από το θόρυβο. και τις προτάσεις που κάνετε εσείς στη γνωμοδότηση σας μπορώ να σας πω ότι μπορώ όλες να τις υπογράψω είναι στόχοι τους οποίους και εγώ θέλω να υπερασπιστώ ως ε, γενικός συζητητής και να τους προωθήσω αλλά δεν ξέρω καθόλου κατά πόσο θα τα καταφέρουμε γιατί είναι τα χέρια μας τόσο δεμένα όπως σας περιέγραψα που δεν ξέρω τι θα βγει. Μπορώ να το πω και εξ ονόματος όλων των συναδέλφων της Επιτροπής ότι τα σημαντικότερα δικά σας μελήματα θα φροντίσουμε να παραμείνουν άθικτα ως προς τα ποσά και να υλοποιηθούν στο ακέραιο. Αλλά ειλικρινά δεν το πολύ πιστεύω. Ούτε μπορώ να σας το υποσχεθώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το σημείο 8 της νομοδότησης, γιατί υπάρχουν πολλοί οργανισμοί στη δική σας ε, καθήλυνα αρμοδιότητα και εγώ δεν είμαι μόνο γενικός ηγητής για τον προϋπολογισμό του 2017, αλλά είμαι και μόνιμος εισηγητής για τους εξωτερικούς οργανισμούς, agencies. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται εκεί. Και εδώ, σε μικρογραφία, αλλά και γενικότερα αντίστοιχα ισχύουν. Δηλαδή αυξάνονται οι ε, προκλήσεις, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες των οργανισμών και μειώνονται τα χρήματα. Θέλω πάρα πολύ να συζητήσουμε τις δυνατότητες ε, που έχουν και στο μέλλον. Να πω κάτι που δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με τον προϋπολογισμό, αλλά με τους οργανισμούς. Θα μπορούσα να φανταστώ σε οργανισμούς που εν μέρει χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία, ας πούμε οργανισμός για τις χημικές ουσίες, θα μπορούσε να αντλήσει περισσότερα κονδύλια από εκεί και να αποσυμφορήσει κάπως τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αξίζει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με την Επιτροπή σας. Ίσως όχι σήμερα έτσι σε τέτοια έκταση. Ας επικεντρωθούμε προς το παρόν στον προπολογισμό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή που ήρθε για να μας ε, παρουσιάσει τις προτεραιότητες για τον προπολογισμό για το 2017. Και όπως είχα πει και προηγουμένως, ε, πρόκειται για μια διαδικασία κάπως αντικανονική, γιατί γίνεται ύστερα, μετά από τα υπόλοιπα. Όπως όλοι γνωρίζετε, τα κλιματικά και περιβαλλοντικά θέματα είναι οριζόντια. Διέπουν όλα τα άλλα και άρα είναι υπό την αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, αλλά στην πραγματικότητα αγγίζουν το, το περιβάλλον σε όλες τις πτυχές και άρα είναι θέματα που απασχολούν όλους. Η Συμφωνία του Παρισιού και όλα όσα έγιναν μετά από αυτήν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, στον προπολογισμό της Ευρώπης. Ε, δεν μπορεί αυτός να μην είναι ευθυγραμμισμένος με τις προτεραιότητες που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επ' αυτού θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή, διότι όλα τα περιβαλλοντικά προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό θα πρέπει να έχουν το ε, την απαραίτητη οικονομική στήριξη αλλά έτσι ώστε να μπορούν πλήρως να εφαρμοστούν όπως γνωρίζει πολύ καλά ο εισηγητής συχνά τα υποχρεώσεις και οι πληρωμές δεν είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και συχνά έχουμε δυσκολία στις πληρωμές που καθυστερούν την εφαρμογή, την εκτέλεση του προπολογισμού και καθιστούν δύσκολη την ε, συντήρηση και την ε, υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Εγώ ήμουν εισηγητής για το προπολογισμό το 2013 και από το 2013 και αλλά και τα υπόλοιπα χρόνια η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, δεν έχει βελτιωθεί. Έχω την εντύπωση λοιπόν πως λοιπόν, είναι απαραίτητο το νέο πολιετές ε, πλαίσιο, η αναθεώρηση δηλαδή αυτού, να λάβει υπόψη αυτές τις δυσκολίες εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Και πήγε προχωρά στη θέματα που εκφράζονται στην γνωμοδότηση. Από τη μια πλευρά έχουμε ένα αίτημα για πλήρη εκτέλεση του προπολογισμού, διατήρηση παράλλακτων των πόρων που προβλέπονται από το PDP ε, για τα προγράμματα που αφορούν αυτή την Επιτροπή, να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε υποχρεώσεις και πληρωμές, έτσι ώστε αυτές οι πολιτικές να μπορούν να εφαρμόσουν και τέλος σε αναφορά στους οργανισμούς. Όπως έκανε και η συγητή, θα πρέπει οι οργανισμοί διάφοροι να μπορούν να ανταποκρίνονται στους υποχρεώσεις που τους έχουν ανατεθεί. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι ε, κάποιοι περιορισμοί, ιδιαίτερα στο προσωπικό, θα εφαρμόζονται ε, αδιακρίτως σε όλους τους οργανισμούς για να μειωθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του προπολογισμού, την εκτέλεση του προπολογισμού. Πολλοί οργανισμοί, όπως είπε ο εισηγητής, και, και εγώ το υπογραμμίζω αυτό, πολλοί οργανισμοί παίρνουν ένα σημαντικό κομμάτι του προπολογισμού από ιδιώτες και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις λειτουργίες τους αν και δεν ζητούν επιπλέον ποσά γιατί έχουν περιορισμούς στο προσωπικό. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο παρανερχόμαστε κάθε χρόνο στη συζήτηση του προπολογισμού και αυτή τη φορά θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Τώρα, από τους Σκιώδης έχουμε τη συνάδελφο για την Μάκη. Πρίγω. Παρακαλώ. Thanks. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, ε, θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο και τον εισηγητή, τον κύριο Γκέιερ. Είμαι αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Γνωρίζω ότι το δημοσιονομικό είναι ιδιαίτερα δύσκολο ε, πρέπει να γίνουν περικοπές, ασκούνται πολλές πιέσεις. Εγώ η, η ίδια ε, προασπίστηκα την ε, τι περικοπέ ε, στο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα, δημοσιονομικά προβλήματα σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα κονδύλια που διαθέτουμε και ενδεχομένως να επινοήσουμε και νέες μεθόδους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους, υπάρχουν διασωτικά προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι αφορά τα δικά μας ζητήματα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, δεν μπορούμε να κάνουμε ε, περικοπές όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή. Ε, δεν μπορούμε να παζαρεύουμε. Σίγουρα τα κονδύλια δεν είναι τεράστια, αλλά πάντοτε υπάρχουν, υπάρχουν. Και πρέπει να τα βρούμε. Ό,τι χρειάζεται πρέπει να το βρούμε. Βέβαια τα κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Αυτό είναι η, η δική μας άποψη. Η Επιτροπή μας επίσης πρέπει να υπογραμμίσει το 20% θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το κλίμα. Αυτό είναι δέσμευσή μας και θα πρέπει να περάσουμε από μια οικονομία άνθρακα σε μια καινούργια οικονομία. Η χρηματοδότηση για αυτούς τους στόχους προφανώς είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ευχαριστώ. Κυρία Κάτεμπακ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαι πολύ αισιόδοξη ότι σε συνεργασία με τον εισηγητή μας θα ε, βρούμε ε, μια λύση, θα έχουμε μια ευρύτατη γνωμοδότηση και μαζί με τον Γιάννη Σαγκάιερ θα προωθήσουμε τα μελήματα του Κοινοβουλίου. Συμφωνώ με την μετα... Ε, προλαλή σας. Στον προϋπολογισμό θα πρέπει να δούμε ότι αυτό που ισχύει σε ένα κρατικό προϋπολογισμό ισχύει και για τον ευρωπαϊκό. Δηλαδή όταν έχουμε επενδύσεις στην υγεία, στην κλιματική αλλαγή, ε, επενδύσεις στραμμένες προς το μέλλον, συνεισφέρουμε στην οικονομία και μακροπρόθεσμα ελαφρύνει το φορολογούμενος αν κάνουμε σωστή πολιτική με το βλέμμα στο μέλλον και πάλι. Δεν είναι δαπάνη αυτό. Μακροπρόθεσμα έχει κέρδος. Και τώρα θα τρέχουμε πάλι να κάνουμε διορθωτικούς και συμπληρωματικούς προπολογισμού. Έχουμε σχέδια ε, παντού και στην κλιματική αλλαγή και όχι μόνο. Ε, θέλουμε ενεργειακή ασφάλεια, θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει ένας τόπος ε, βιομηχανικής παραγωγής και οικονομικής παραγωγής για να γίνει αυτό πρέπει να κάνουμε τις σωστές κινήσεις και είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε να το κάνουμε ε, για το 2017 και να ανταποκριθούμε και στις απαιτήσει και στις προσδοκίες των πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Κονέτσνα. Δεν θα επαναλάβω οτιδήποτε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή της Επιτροπής Προπολογισμών Έχουμε αφιερώσει πολύ χρόνο σε αυτό το θέμα. Έχουμε όλο και περισσότερα δημοσιονομικά προβλήματα και όλο και περισσότερα αρμοδιότητες, <clears throat> καθήκοντα, τα οποία πρέπει να χρηματοδοθούν με όλο και μικρότερους πόρους. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα. Έχουμε ανάγκες προϋπολογισμού, δημοσιονομικές ανάγκες. Από την άλλη μεριά είναι περιορισμένοι οι πόροι μας. Ε, έχουμε υποχρεωτικές δαπάνες, ανελαστικές δαπάνες, ε, είναι πολύ δύσκολο ε, να τα βγάλουμε πέρα, πλην όμως χαίρομαι που ο εισηγητής, τουλάχιστον ό,τι αφορά τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταφέρνει να τους εξασφαλίσει αρκετούς πόρους ώστε να φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά τους. Γιατί χρειαζόμαστε ειδικευμένες υπηρεσίες, αυτές έχουν εμπειρογνώμονες, οι εμπειρογνώμονες πρέπει να πληρώνονται γιατί αλλιώς δεν θα καταφέρουμε να παίρνουμε τις σωστές πολιτικές αποφάσεις. Έχουμε έλλειψη πόρων στο δίκτυο Natura 2000. Έχουμε συνεχείς μειώσεις των επιχορηγήσεων των πόρων κάτι που μας οδηγεί στο να μην μπορούμε να ε, είμαστε συνεπείς με τις υποσχέσεις μας. Και αυτό μας ε, το επισημαίνουν τα κράτη-μέλη. Θέλουμε όλο και περισσότερες ζώνες να εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 και από την άλλη μεριά μειώνουμε τους πόρους του δικτύου. Συνεχώς. Ας μην το ξεχάσουμε λοιπόν αυτό το θέμα. Γιατί ένα πράγμα είναι τι γράφουν τα χαρτιά και ένα διαφορετικό είναι ότι γίνεται στην πράξη στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει ο προπολογισμό να βοηθάει τα κράτη-μέλη. Και για την περίπτωση Natura 2000 πρέπει να βρούμε μια λύση. Μέσω του προπολογισμού. Για μας είναι προτεραιότητα. Στα χαρτιά είναι προτεραιότητα όλων, αλλά μερικέ φορέ έχουμε προβλήματα πόρων και χρηματοδότηση. Βιοπικιλότητα. Η βιοπικιλότητα επίση πολύ σημαντική. Θα υποβάλουμε και συγκεκριμένη τροπολογία για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή της Επιτροπής Προπολογισμών και παρόλο ότι δεν είμαστε θετικοί σε όλα, θα συνεισφέρουμε στην βελτίωση του τελικού κειμένου για να πετύχουμε και τους στόχους του 2017. Κύριε Μελλέρ, ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Καλή έκθεση. Ε, θα ήθελα να τονίσω εδώ κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Στην παράγραφο 8 αναφέρει ο συγητής στους οργανισμούς Ακριβώς η οικονομική κατάσταση των οργανισμών είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε. Ε, τους δε τελευταίους μήνες στη συζήτηση για το γλυφοσάτ και τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς είδαμε ε, να διακυβεύεται η ανεξαρτησία ε, και η ε, αξιοπιστία ιδιαίτερα του ΕΦΣΑ. Ο κόσμος το αμφισβητεί αυτό μαζικά. Τώρα, άμα θέλετε να δώσετε λιγότερα χρήματα ακόμα στους οργανισμούς για να τα παίρνουν περισσότερο από τους ιδιώτες, δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ως πολιτικοί πρέπει να έχουμε τεκμηριωμένη ενημέρωση με στοιχεία για να παίρνουμε σωστές ε, πολιτικές αποφάσεις. Και εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι, δεν θα, ότι θα είχε νόημα ε, κάτι τέτοιο. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο, να δώσουμε εμείς περισσότερα χρήματα για να είναι δεδομένη η ανεξαρτησία της επιστήμης. Αυτός ε, είναι ο πιο σωστός δρόμος και ο πιο ευγνώμων και ο λιγότερο αχάριστος δηλαδή. Ε, προς τους ανθρώπους αυτούς που μας βοηθούν να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Είναι λάθος ότι θα πρέπει να βγούμε από τον προπολογισμό τους και να τους ρίξουμε στην αγκαλιά ε, της ε, βιομηχανίας. Ευχαριστώ, η κυρία Κροστέτ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομη θα είμαι. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή και είναι λυπηρό πραγματικά επειδή έχουν στη Βρετανία δημοψήφισμα εμείς να καθυστερούμε στις εργασίες μας. Δεν θα ήταν καλύτερο να επιδεικνύει την προθυμία της η Ευρώπη να προχωράει όλο και περισσότερο. Αυτό είναι ομολογία αδυναμίας και είναι κρίμα. Συμφωνώ πάντως και με τον εισηγητή και με τους συναδέλφους. Έχει μεγάλη σημασία να υπερασπιστούμε τον προπολογισμό των οργανισμών και μεταξύ αυτών με τις οποίες, εκείνες με τις οποίες συνεργαζόμαστε περισσότερο του ζητάμε όλο και περισσότερα πράγματα να κάνουν και μας το λένε κάθε φορά ότι είναι πολύ πιο δύσκολο πια να απαντήσουν στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί δεν δίνανται. Τουλάχιστον να μην περικοπεί ο προπολογισμό του ζητάνε, όχι αύξηση. Αφήστε που χρειάζεται κάποια μικρή αύξηση αν γίνεται να προσπαθήσουμε. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο να λειτουργήσουν οι οργανισμοί με τα χρήματα που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή. Ας δείξουμε λοιπόν την προθυμία μας και τη βούλησή μας να μην την πληρώσει ο προπολογισμό. Γιατί δηλαδή επειδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρές και βαριές κρίσεις θα πρέπει κάθε φορά να περικόπτουμε τα χρήματα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και έτσι και αλλιώς γελίος σε σχέση με ε, τα όσα καλούμαστε να κάνουμε. Οπότε θα ήταν καλύτερο και προτιμότερο να δείξουμε στα κράτη-μέλη ότι διαφωνούμε με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται αυτά τα θέματα και θέλουν να ε, κυβερνούν και να δικούν την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο. Όχι. Οπότε να δώσω μέσα το λόγο στο Γενικό Εισηγητή μας, τον κύριο Γκάιερ, για να κλείσει τη συζήτηση αυτή. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Μερικά σημεία να συνοψίσω μόνο. Πρώτον, διαδικαστικά. Είναι πραγματικά λυπηρό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα καθυστερεί, ανέβαλε κατά τέσσερις εβδομάδες τη δημοσίευση του σχεδίου προϋπολογισμού. Αλλά με αυτό δεν έχουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεγάλα προβλήματα θα γλιτώσουμε και μια έκθεση. Συνήθως στη διαδικασία αυτή, στο επόμενο βήμα προβλέπεται συζήτηση για την εντολή, για το τριμερή διάλογο, με το Συμβούλιο και την Επιτροπή δηλαδή, για θέματα δημοσιονομικά. Την έκθεση αυτή, για λόγους χρονικούς, δεν θα μπορέσουμε να την υποβάλουμε, γιατί κανονικά αυτή κατατίθεται πριν ε, τις δεκοπέ. Αν πάρουμε τέλη Ιουνίου τώρα το σχέδιο προπολογισμού, Χαιρετίσματα. Δεν φτάνει ο χρόνος. Μένα δεν με πειράζει, εντάξει, μια έκθεση λιγότερη. Με το όνομά μου δεν χάλασε και ο κόσμος. Από τις νομιμοδοτήσεις των επιμέρους επιτροπών θα χτίσουμε μια εντολή. Είναι μια διαδικασία που έχει δοκιμαστεί, γιατί και το 2014 το ξαναζήσαμε, επειδή είχαμε ευρωεκλογέ, ήταν πάλι ε, πιεσμένα τα χρονοδιαγράμματα και είχαμε και μια πιο σύντομη διαδικασία για τις ευρωεκλογέ. Ξέρετε ότι οι κοινοβουλευτικές εργασίες σταματούν έξι εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογέ. Τότε φταίγαμε εμείς, τώρα φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτός που θα έχει πρόβλημα είναι η Σλοβακική Προεδρία, που έτσι κι αλλιώς έχει έναν εκνευρισμό και ένα άγχος, γιατί είναι η πρώτη Προεδρία των Σλοβάκων. Εάν τους πιέσουμε και χρονικά στον προπολογισμό, θα πελαγώσουν οι άνθρωποι. Εμείς στο Κοινοβούλιο, επαναλαμβάνω, τα έχουμε αυτά υπό έλεγχο. Θα ήθελα να ε, καθισκάσω λίγο τον συνάδελφο Λαβία για τις πληρωμές σε σχέση με την ανάληψη υποχρεώσεων. Εμείς γνωριζόμαστε από καιρό είμαστε στο, στο, στην Επιτροπή προπολογισμού. Με ε, το νέο πλαίσιο, το PDP, έχουμε καινούρια χρήματα και κάπως η κατάσταση αυτή έχει εξισορροπηθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να εξοφλεί λογαριασμούς. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, μια κουβέρτα που φτάνει μέχρι το λαιμό. Την τραβάς και σκεπάζει το λαιμό σου, βγαίνουν τα, πέδια, ε, τα πόδια απ' έξω και κρεώνουν τα πόδια σου. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι να τραβάς την κουβέρτα πάνω κάτω, <laughs> αλλά να βρεις μια κουβέρτα που να καλύπτει ε, όλο το σώμα. Και να δούμε ε, γιατί μέχρι να τελειώσει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα έχουμε λεφτά για τις πληρωμές. Αλλά θα έχουμε λάβει άλλες υποχρεώσεις και αυτού και από την αρχή. Αυτό το πρόβλημα του προπολογισμού είναι διαρθρωτικό και θα πρέπει να λυθεί εκεί. Το συζητούμε με πάσα ευκαιρία με το Συμβούλιο και στην αναθεώρηση θα τα πούμε πάλι. Αλλά, και έρχομαι εδώ στο δεύτερο θέμα που θίξατε, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυστυχώς και είναι από τα λίγα μειονεκτήματα της τη της Λισαβόνας, δεν έχουμε την ισχύ και την εξουσία που είχαμε στο παρελθόν γιατί χάσαμε τη δεύτερη ανάγνωση. Δηλαδή, θα πρέπει να συμφωνήσουμε το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και αυτό είναι το πρόβλημα. Και για να το πω λίγο άκομψα, έχουμε ε, μία πυρηνική βόμβα ε, στο τουλάπι μας ε, να απορρίψουμε τον προϋπολογισμό ε, και ε, τι σημαίνει αυτό ότι θα συνεχιστεί ο προϋπολογισμός του 2016 και όπως το λέει η τεχνική γλώσσα είναι τα προσωρινά 12 τιμόρια κάθε χρόνο μεταφέρει στον ε, αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Γίνεται και αυτό αλλά θα πρέπει να ακούσουμε τι λένε οι συνάδελφοι από τις επιτροπές που έχουν περισσότερα χρήματα ε, και έχουν να καλύψουν ε, την ε, πολιτική ευθύνη. Περιφερειακή πολιτική, γεωργία, έρευνα. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν είναι από πολλά κονδύλια, αλλά υπάρχουν πιο πολλές επιτροπές που χειρίζονται άλλα προγράμματα. Ας πούμε, τα ΕΣΠΑ, πώς θα τρέξουν αν πάμε σε 12 τιμόρια. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ισχύ μόνο στο βαθμό που είμαστε ενωμένοι και μπορούμε να ενώσουμε μεγάλη πλειοψηφία σε ένα πολιτικό εγχείρημα. Και μόνο ε, ε, αρκεί να αναφερθεί η απόρριψη του προπολογισμού για να διχαστούμε. Όλες οι επιτροπές γκρινιάζουν, δεν μας φτάνουν τα λεφτά και αυτές οι επιτροπές που σας ανέφερα λένε ότι συμφωνούν να απορρίψουμε τον προπολογισμό. Ναι, αλλά τότε αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί ε, θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να συγκρουστούμε. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί. Ε, στις προηγούμενες συζητήσεις ε, για τον προϋπολογισμό είχαμε μεγάλες δυσκολίες. Στην ε, Λουξεμβουριανή Προεδρία όμως πήγαν πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι κατάφερε η Προεδρία να ε, λύσει τις διαφορές που είχε το Συμβούλιο η Αντιπρόεδρος κυρία Γεωργίευα, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολύ εύστοχα είχε πει το εξή. Ότι στο Συμβούλιο είναι τρεις οι ομάδες. Αυτά που σας λέω τα ανέφερε κυρία Γεωργίευα, είναι δική της οι χαρακτηρισμοί. Είναι οι φίλοι της γεωργικής πολιτικής, οι φίλοι των εκπτώσεων και οι φίλοι της συνοχής. Και αυτές οι τρεις ομάδες διαφωνούν απολύτως μεταξύ τους στο Συμβούλιο, αλλά κάπου καταφέρνουν να φέρουν μια κοινή θέση που πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς λοιπόν οι φίλοι των εκπτώσεων, που είναι και η πατρίδα μου μέσα σε αυτές τις χώρες, ε, αγωνίζονται πάρα πολύ να περικόψουν τις πληρωμές. Γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πόσο θα επιβαρυνθεί συγκεκριμένα ο κρατικός προϋπολογισμός. Πόσα λεφτά θα πρέπει να στείλω στις Βρυξέλλες και όσο λιγότερα τόσο καλύτερα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε το εξή τώρα. Πολλά κράτη-μέλη θα προσπαθήσουν να κάνουν περικοπές στις πληρωμές και θέλω από τώρα να δεσμευτώ ενώπιόν σας ότι θα το προσέξω στην κατηγορία 3 και τα προγράμματα της ΕΝΒΗ δεν θα γίνουν και άλλες περικοπές. Υπάρχει ένα μικρό περιθώριο στην κατηγορία 2. Το live δεν απειλείται κατά με, αλλά έχουν μια μανία να περικόπτουν στις πληρωμές και ψάχνουν για νέα θύματα που ελπίζω να μην είναι τα περιβαλλοντικά προγράμματα. Ε, κυρία Μίλλερ, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Να το πω πιο συγκεκριμένα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να έρχονται περισσότερα ιδιωτικά χρήματα στους οργανισμούς, από τη βιομηχανία δηλαδή. Δεν θέλω να προσελκύσω περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις της βιομηχανίας. Αφήστε που δεν υπάρχει υποχρεωτική ε, σύνδεση ε, πληρωμών των κρατών μελών και ανεξαρτησίας των οργανισμών. Δεν σημαίνει ότι επειδή χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη είναι ανεξάρτητα. Έχουμε ζήσει και στο παρελθόν καταστάσεις, ε, ας πούμε, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ε, με κάποιες ε, μελέτες και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων που γνώρισαν τεράστια αμφισβήτηση και έγινε και αλλαγή. Το ξέρω πολύ καλά τον διευθυντή της ΕΜΑ του ΕΟΦ και το, γιατί δούλευε στο κοινοβούλιο ήταν διοικητικός υπάλληλος και μου είπε Γιάννης μπορείς να δεις τι γίνεται με στα πανεπιστήμια. Μπορείς να βρεις σε όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης ένα καθηγητή φαρμακευτικής που να μην έχει δουλέψει ποτέ την τελευταία τριετία για φαρμακοβιομηχανία. Γιατί είναι σχετικό το θέμα αυτό της ανεξαρτησίας των εμπειρογνωμόνων. Πού να τον βρούμε αυτόν που δεν έχει συνεργαστεί με τη βιομηχανία. Μπορεί να είναι πολύ ωραία πρόθεση, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ακριβώς ε, χρειάζονται επιστημονική υποστήριξη και αν τους κόψουμε αυτούς δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν τίποτα εμπειρογνώμονες και επιστήμονες ανεξάρτητοι που να μην ε, ε, συνεργάζονται. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ έδρα σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που να λέει ότι όχι, εγώ δεν θέλω τέτοια πράγματα. Θέλω να παραμείνω αγνός και αλόβητος και να μην ασχολούμαι με αυτά. Ε, είμαι εμπειρογνώμων για Ευρωπαϊκό Οργανισμό, άρα ε, ε, απορρίπτω ένα ερευνητικό πρόγραμμα της βιομηχανίας. Δεν έχει γεννηθεί αυτός ο άνθρωπος ακόμα. Λοιπόν, οι ε, οργανισμοί αυτοί παρέχουν υπηρεσίες στη βιομηχανία. Ελέγχουν μια ουσία, ελέγχουν ένα παρασκεύασμα, καταγράφουν, κατοκυρώνουν ένα προϊόν, δεν ξέρω, κάποια αρμοδιότητα που τους έχει αναθέσει η Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Και η ε, βιομηχανία πληρώνει ένα τέλος για να γίνει αυτό. Μήπως μπορούμε να αυξήσουμε αυτό το τέλος, ας πούμε, για να συνεισφέρει αυτό στη χρηματοδότηση του οργανισμού για να ελαφρυνθεί κάποιος, ο, κάπως ο ευρωπαϊκός προπολογισμό. Και ενδεχομένως να μπορέσουν να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό, συμφωνώ απολύτως, ή να αλλάξουν τη δουλειά τους κάπως. Εγώ θα πρέπει να ασχοληθώ με την εξή κατάσταση. Από τη μια μου λένε οργανισμοί, κύριε Γκάιερ, αυξάνονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες και έχουμε εξαντλήσει τα όρια μας. Και από την άλλη, Έγινε αυτή η τρομερή συμφωνία το 2013 ε, σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ και παντού και στους οργανισμούς να γίνουν περικοπές στο προσωπικό κατά 5%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς να πω, δεν έχει αθροίσει όλες τις υπηρεσίες και όλους τους οργανισμούς μαζί και, και είπε από αυτό το πουλ θα κοπούν 5%. Όχι, σε κάθε ξεχωριστή υπηρεσία θα κόβεται 5%. Υπάρχουν και οργανισμοί που δεν χάνουν 5% αλλά 10% ε, για να πηγαίνουν ε, οι, πάλι, οι θέσεις μάλλον στο redeployment pool γιατί συνενώνονται οι θέσεις που χειρεύουν. Ξέρετε στα κράτη-μέλη πόσο δημοφιλές είναι όταν ζητάς να στείλουν περισσότερα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί να δείτε πειρά ομαδών. Στη Γερμανία, αν βγεις και πεις θέλουμε περισσότερα λεφτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ δεν φοβάμαι να συνεχίσω να το κάνω, γιατί ξέρω ότι έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι οφείλει να κάνει βάσει των συνθηκών και θα πρέπει να κάνει τη δουλειά τη. Οπότε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κανονίσουν την πορεία του. Είτε θα στείλουν περισσότερα λεφτά, είτε θα καταλήξουν στου ιδίου πόρου για να συμφωνήσουν ποιοι θα είναι αυτοί. Γι' αυτό μίλησα για τέλη, ας πούμε, ε, στους οργανισμούς από την ε, ιδιωτική ε, βιομηχανία και μπορούν να προέρθουν από εκεί χρήματα για τον προπολογισμό. Αυτή είναι άλλη συζήτηση όμως. Μπορούμε να την κάνουμε κυρία Μιούλερ. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει και είμαι στη διάθεσή σας πάντα. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Good afternoon, everybody. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ έχω μόνο ένα καθήκον σε σχέση με αυτόν τον φάκελο. Να σας ενημερώσω για το χρονοδιάγραμμα για την ε, γνωμοδότηση για την εντολή για το τριμερή διάλογο. Ε, η προθεσμία είναι η 31η Μαΐου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΝΒΗ στις 21 Ιουνίου. Ολομέλεια θα ψηφίσει τον Ιούλιο. 4 με 7 Ιουλίου στην Ολομέλεια. Και στην Επιτροπή Προπολογισμού η παρουσίαση του σχεδίου έκθεση προβλέπεται για τι 15-16 ε, Ιουνίου και η Επιτροπή Προπολογισμού θα ψηφίσει στι 30 ε, Ιουνίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ κύριε Γκάιερε που ήσασταν εδώ με την Επιτροπή ΕΝΒΗ και για τη συμβολή σας και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερή διάταξη, που είναι η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Αξιολόγηση Εφαρμογής του Κανονισμού σχετικά με υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με το τρόφιμα. Και εδώ θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση μιας μελέτης για 10 λεπτά. Να ζητήσω από την Εκατερίνα Καραφίλοβα από την ε, Επιτροπή να μας κάνει αυτήν την ε, παρουσίαση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη. Ονομάζομαι Εκατερίνα Καραμφίλοβα. Ε, εργάζομαι στο EPRS. Ε, το κέντρο, η υπηρεσία έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος μας είναι να, στηρίξουμε, να στηρίζουμε το έργο των επιτροπών και ε, να ε, κρίνουμε αξιολογίες εφαρμογής των ευρωπαϊκών κειμένων. Ορισμένες από τις δημοσιεύσεις μας βλέπετε στην οθόνη. Ε, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα των υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ε, η μελέτη μας έχει ως στόχο να προετοιμάσει συζήτηση για το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, αξιολογούμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής του κανονισμού 1935 του 2004 που καθορίζει συγκεκριμένους στόχους και απαιτήσεις για τα υλικά αυτά. αντιπροσωπεύει μια έρευνα που κάναμε εμείς ε, ε, μεταξύ Δεκεμβρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2016 με τους βασικούς ενδιαφερόμενους. Ε, βασικοί ενδιαφερόμενοι είναι επιχειρήσει, κράτη-μέλη, καταναλωτέ, μη κυβερνητικέ οργανώσει και ερευνητέ. Και τα 28 κράτη-μέλη έλαβαν, έλαβαν μέρο μέσω των αρμόδιων αρχών του, όπω επίση η ΕΦΣΑ και η Επιτροπή. Λάβαμε συνολικά 61 συνεισφορές από ενδιαφερόμενους. Οπότε είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Πολύ αντιπροσωπευτικό. Ε, εκ μέρους της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν. Συλλέξαμε στοιχεία μέσω ενός ε, ερωτηματολογίου που έλεγξε το πώς εφαρμόζεται ε, ο κανονισμός σε σύγκριση με τα όσα προβλέπει για παράδειγμα συνέπεια σε σχε, σχετική σχέση με το, το κείμενο προσθέμενη αξία, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συμπληρωματικότητα, χρησιμότητα. Ε, η μελέτη εντοπίζει συγκεκριμένε τάσει σε ό,τι αφορά την αντίληψη που έχουμε για την εφαρμογή του διάφορου ενδιαφερόμενοι. Τα, τα συμπεράσματα είναι ότι υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, ένα πρόβλημα με το νομικό πλαίσιο της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον υπάρχει ένα πρόβλημα με την εφαρμογή των κανόνων. Να σας, πω, να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Ως γενική τάση, οι ενδιαφορμοί θεωρούν ότι το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή δεν είναι πλήρες. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για ορισμένα πολύ χρησιμοποιούμενα υλικά. Για ποιο λόγο, γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό οι ε, ουσίες που μεταναστεύουν από το υλικό στο φαγητό δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή να αλλοιώνουν τις ίδιες τροφές. Πρόκειται για ένα όρο που αφορά όλα τα υλικά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Από, 17, από τα 17 υλικά τα οποία αναγράφονται στο παράρτημα του κονισμού, ε, υιοθετήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται και πρέπει να εφαρμόζονται. Οπότε αν δεν υπάρχουν ειδικά μέτρα για συγκεκριμένα υλικά, επηρεάζεται η εφαρμογή του κανονισμού. Ειδικά μέτρα δεν έχουν υιοθετηθεί για όλα τα υλικά και σε αυτήν την περίπτωση τα κράτη-μέλη έχουν, μπορούσαν να υιοθετήσουν ειδικά του εθνικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή έχουν υιοθετηθεί ειδικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέσσερα, για τέσσερα υλικά. Πλαστικά, κεραμικά, ε, αναγεννημένη κυταρίνη και ευφυή και ενεργά υλικά. 13 άλλα υλικά του καταλόγου δεν έχουν τύχει εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Ορισμένα κράτη-μέλη βέβαια έχουν υιοθετήσει σε εθνικό επίπεδο μέτρα, ειδικά μέτρα για αυτά τα υλικά. Και εκεί, και από εκεί πηγάζει το πρόβλημα. Γενικά, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι ε, για τα υλικά τα οποία δεν, δεν έχει γίνει εναρμόνιση, ε, δεν είναι δυνατόν να ε, συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες που υφίστανται. Γιατί? Γιατί οι αγορές για αυτά υλικά καταστρέφονται εξαιτία της ύπαρξης διαφορετικών κανόνων σε διάφορα, σε διάφορα κράτη-μέλη. Γι' αυτό το λόγο η έλλειψη ευρωπαϊκών κανόνων για ορισμένα υλικά έχει αρνητική επίδραση στις αγορές. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα όπως τα αναφέρουν οι ενδιαφερόμενοι οι αρνητικές επιπτώσεις μέσω φραγμών στην εσωτερική αγορά, ε, δεν γίνεται εξασφάλιση εννέων κανόνων ασφάλειας, αύξηση των κανόν, των, του κόστου συμμόρφωσης, γραφειοκρατικά προβλήματα εξαιτία διαφορετικών συστημάτων αδειοδότησης, ε, μείωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, μείωση της, των ευκαιριών βελτίωσης των τροφίμων μέσω καινοτομίας για όλους αυτούς τους λόγους ε, πολύ ενδιαφερόμενοι ζητούν να υιοθετηθούν ειδικοί κανόνες και για τα μη εναρμονισμένα υλικά. Όπως βλέπετε σε αυτό το πίνακα, ε, το χαρτί και το χαρτόνι ε, είναι αυτό που πιο πολύ χρειάζεται εναρμόνιση. 62% των ενδιαφερομένων το ζήτησαν. Σε ό,τι αφορά το εύρος της εναρμόνισης, πρόκειψαν δύο συστάσεις. Πρώτον, ειδικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να ε, βασίζονται σε ε, ομοιόμορφους κανόνες ε, δοκιμών, έτσι ώστε και οι αρμόδιες αρχές και οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να κάνουν τις δοκιμές με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, αυτή η προδιαγραφή θα πρέπει να είναι ειδική για κάθε υλικό, γιατί κάθε υλικό έχει τις ιδιαιτερότητες του. Θα πρέπει να αποφύγουμε τη σημερινή κατάσταση όπου τα μη εναρμονισμένα υλικά δοκιμάζονται με μεθόδους οι οποίες έχουν επινοηθεί για τα εναρμονισμένα υλικά. Αυτό οδηγεί σε αμφισβητούμενα αποτελέσματα. Οι ενδιαφερόμενοι επίσης επιμένουν ότι η υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων σε ευρωπαϊκό πεδίο θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και η απόφαση θα πρέπει να ε, προσαρμόζεται σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα. Επίσης, συστήνουν καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους ε, παίκτες που ε, κατέχουν τη γνώση, που έχουν τεχνογνωσία, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως των ουσιών που έχουν ε, προσθεθεί ε, μη σκοπίμως και άλλου τύπου προβλήματα. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, τα προβλήματα που αναφέρθηκαν έχουν σχέση με την ίχνη λασιμότητα, την, την, τα έγγραφα τα οποία τα αποδεκτικά της συμμόρφωσης και τους ελέγχους. Οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι η δηλώση συμμόρφωση είναι σημαντική σε ό,τι αφορά την χνηλασιμότητα ε, για τα υλικά που εισάγονται και για τα υλικά που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι ότι ε, είναι θέμα διαθεσιμότητας τέτοιων ε, δηλώσεων αλλά και ε, αξιοπιστίας τους και ποιότητας αυτών των δηλώσεων. Ε, οι δηλώσει που είναι χαμηλή ποιότητα δυσκολεύουν την ιχνηλασιμότητα. Γι' αυτό το λόγο συστήνουν πρώτον ε, κατάρτιση, ειδική κατάρτιση και για τις αρμόδιες αρχές και για τους επιχείρησει, έτσι ώστε να βελτιωθεί η συμμόρφωση αφενός και η επιβολή του αφετέρου. Δεύτερον, ε, να γίνουν προσπάθειες έτσι ώστε να βελτιωθεί η χνηλασιμότητα των εισαγόμενων υλικών και τρίτον, η εισαγωγή ε, υποχρέωσης ε, ε, ταυτοποίησης των υλικών αυτών. Η έλεγχη αναφέρεται ότι δεν γίνονται με την ίδια σοβαρότητα σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν είναι σωστό. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για αυτό το θέμα δεν είναι αρκετές ώστε να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Θα πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ε, ελεγκτικές ε, δραστηριότητες, τη συχνότητά τους, τους ελέγχους των δηλώσεων συμμόρφωσης και τους ελέγχους εισαγωγών. Θα πρέπει να γίνει μια χαρτογράφηση των αναγκών προκειμένου να αναπτύξουμε και άλλα ε, νομικά εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό ζητούν οι ενδιαφερόμενοι. Ε, εδώ βλέπετε μια σύνοψη της, ε, της αξιολόγησης ε, εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι οι κανόνες πληρούνται καλύτερα για τους, μάλλον οι στόχοι περί και ασφάλειας τηρούνται περισσότερο για τα εναρμονισμένα υλικά. Και μάλιστα ε, τα ενορισμένα υλικά έχουν δώσει και προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους. Ευχαριστώ πολύ. Και μετά την ε, παρεπόμενη παρουσίαση της ε, έκθεσης θα απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Σάλντε Μόζε. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ για αυτή την εξαιρετική εισήγηση. Αυτή η μελέτη με βοήθησε πολύ σήμερα, γιατί πολλά από τα συμπεράσματα είναι συμπεράσματα που και εγώ η ίδια έχω περιλάβει σε αυτή την έκθεση. Νομίζω πως είναι σημαντικό όταν ε, προβαίνουμε σε συστάσεις σε αυτό το τομέα να βασιζόμαστε σε στοιχεία και όχι σε ε, επιθυμίες. Περί πρόκειται. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ισίωση νομοθεσία αποτελεί μια καλή βάση για τη ρύθμιση των προϊόντων που προορίζονται, των υλικών, συγγνώμη, που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Υπάρχουν όμως κάποιες ελλείψεις ε, ιδιαίτερα ε, για μια σειρά ε, υλικών. Ιδιαίτερα όσον αφορά το, την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε την έκθεση αυτή και γι' αυτό και έχω προβεί σε κάποιες συστάσεις εδώ, μια σειρά συστάσεων. Τις λεπτομέρειες θα τις δείτε στην έκθεση. Καταρχάς, θα ήθελα να ζητήσουμε από την Κομισιόν να λάβει περισσότερα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε και για περισσότερα υλικά και ουσίες όπως το χαρτόνι, το χαρτί και η επεξεργασία της επιφάνειας του χαρτιού και του χαρτονιού αλλά επίσης και για το μελάνι που χρησιμοποιείται. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά ε, εταιριών που ζητούν το ίδιο πράγμα και νομίζω ότι εκεί έγινε το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η βασική μου λοιπόν σύσταση, περισσότερα ειδικά μέτρα σε κάθε επίπεδο ώστε να εναρμονιστούν οι ε, διάφορες διατάξεις για τα διάφορα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Άλλη πτυχή είναι η ασφάλεια. Πρέπει η ασφάλεια να ε, είναι εγγυημένη και γι' αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να εξετάσουμε περισσότερο το ρόλο της ε, υπηρεσίας του οργανισμού για την ασφάλεια των τροφίμων. Θα πρέπει δηλαδή να έχει περισσότερους πόρους αυτός ο οργανισμός. Εάν ζητά κανείς ιδιαίτερα περισσότερους πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτό φυσιολογικό. Εάν ζητάτε περισσότερο έρευνε, ε, τότε σημαίνει ότι το ζητάτε από τον αυτόν τον οργανισμό της ασφάλειας για τα τρόφιμα. Όμως θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε αυτός ο οργανισμός να έχει και την κατάλληλη εντολή για να ελέγξει την ασφάλεια αυτών των υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Όλο ένα και περισσότερο βλέπουμε ότι τα κρατημέλη παρατηρούν την ύπαρξη ενδοκρινικών διαταρακτών σε αυτά τα υλικά και γι' αυτό ε, φυσικά είναι προβληματικό. Γι' αυτό και θα πρέπει ο οργανισμός για την ασφάλεια των τροφίμων θα πρέπει όντως να ασχοληθεί με το ζήτημα τόσο όσον αφορά κοκτέιλ υλικών όσον αφορά και ε, τις ε, πολλαπλές ε, επιπτώσεις ή τις, τις επιπτώσεις σώρευσης τέτοιων υλικών. Ε, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι χρειάζονται προτάσεις αλλά και προτάσεις αλλά και διατάξεις για τον έλεγχο. Πώς λειτουργούν οι έλεγχοι σε, αυτός, το, σε αυτά τα υλικά. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Πρέπει να εναρμονιστούν τα πράγματα πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Και εδώ νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι η εγγυήτρια για την εναρμόνιση των ελέγχων και να μεριμνήσει ώστε να υπάρχει και καταρτισμένο προσωπικό που θα προβαίνει σε αυτούς τους ελέγχους. Τώρα, επίσης η ανείχνευση και η πρόληψη είναι σημαντική. Θα πρέπει να μπορούν να, ε, τα κράτη-μέλη να βρίσκονται σε επαφή και να προβαίνουν στις κατάλληλους προληπτικούς ελέγχους. Κύριε Πρόεδρε, περιοριζόμαστε στο μέγεθος της έκθεσης που συντάσσουμε, γι' αυτό και δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω όλα όσα θα επιθυμούσα στην έκθεση αυτή. Θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς, για παράδειγμα, θα μπορέσουμε να καλύψουμε το θέμα της σχέσης ανάμεσα ε, στα υλικά επαφής και την ε, κυκλική οικονομία. Δεν θα πρέπει οι ρυθμίσεις για τα υλικά επαφής να μας εμποδίσουν να ε, στήσουμε την κυκλική οικονομία. Φυσικά θα γίνουν προσθήκες μέσω τροπολογιών που αναμφίβολα θα εμπλουτίσουν την έκθεσή μου. Η νομοθεσία αυτή λοιπόν είναι μια καλή βάση, αλλά υπάρχει τρόπος να βελτιωθεί ακόμη περισσότερη κατάσταση μέσω ειδικών βελτιώσεων στο επίπεδο των ελέγχων των ε, εξετάσεων αλλά και ε, της εντολής ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στο Τρόφιμα. Χαίρομαι που συνεργάζομαι με τους κοιόδης εισηγητές ε, στο θέμα αυτό και να τους ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Μας μένουν μόλις λίγες εβδομάδες για να καταθέσουμε τροπολογίες και να κάνουμε μια πλούσια συζήτηση και σας ευχαριστώ εκ των περιττέρων για τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Αρχίζουμε λοιπόν στις σκοτωσυγητές. Κύριε Κολλάν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να αρχίσω την παρουσίασή μου με μια ρητή ευχαριστία προς την εισηγήτρια την Κρίστελ Σάλτεβος. Ήταν υποδειγματική συνεργασία από πολύ πρώιμο στάδιο. Συζήτηση, κοινέ εκδηλώσεις, πάντα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε αν βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο ή όχι. Θέλω επίσης ρητά να ευχαριστήσω και την υπηρεσία του Κοινοβουλίου για τη μελέτη, ε, ακριβώς ε, αυτά τα θέματα που μας απασχολούν φύγει και εξετάζει ε, ερωτήσεις που είχαμε και οι ίδιοι. Θα ήθελα όμως ε, να απευθυνθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πω ρητά ότι λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχουμε ακόμα την ε, μελέτη του κοινού κέντρου ερευνών. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για τη συζήτηση. Γιατί καθυστερεί αυτή. Μερικές σύντομες παρατηρήσεις, ακούσαμε πολλά έχουμε τέσσερα εναρμονισμένα μέτρα και 13 μη εναρμονισμένα. Από όλα αυτά που άκουσα, ακριβώς στα μη εναρμονισμένα μέτρα, όπως μας παρουσιάσατε, είναι οι μεγάλες δυσκολίες. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν βρει δικές τους λύσεις για αυτά τα προϊόντα, ας πούμε Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία ε, και σε άλλες ε, περιπτώσεις ε, ε, για τα χρώματα και για τις επιστρώσεις όπως και στην Ελλάδα. Εκεί που δεν υπάρχει εναρμόνιση θα πρέπει κανονικά να βρίσκει εφαρμογή η αρχή της αμοιβαία αναγνώρισης. δεν ξέρω αν σας κατάλαβα καλά, θα μπορούσατε να μου απαντήσετε. δεν, λειτουργεί επαρκώ αυτή η αρχή τη αμοιβαία αναγνώριση και θα παρακαλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιληφθεί ε, και να τοποθετηθεί επί του θέματο. Αν λοιπόν δεν λειτουργεί αμοιβαία αναγνώριση, τι γίνεται με αυτά τα 13 μέτρα που δεν είναι αρμονισμένα. Χρειάζεται εναρμόνιση. Ε, Ποιε είναι οι προτεραιότητες ε, ω προ τι ουσίε και τι ομάδε. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καθοδήγηση υπάρχουν μέτρα εθνικά, όπως στη Γερμανία, συστάσεις ε, του ε, Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου για ε, εκτίμηση του κινδύνου ή γιατί γίνεται με τις μελάνες, τα χημικά. Πάντως οι λύσεις όποιες και να είναι θα πρέπει να είναι κοντά στην πρακτική και εφαρμόσιμες και να μην το παρακάνουμε και να μην υπερβάλλουμε. Στις προτάσεις για το πλαστικό βλέπουμε ε, ότι είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένες, πάρα πολύ λεπτομερείς και με χρονοδιαγράμματα. Και το θέμα είναι τι μπορεί να περιλαμβάνει μια συσκευασία ή ε, ένα μαχαιροπύρουν ή άλλα σκεύη. Έχω κάποιες προτάσεις, θα κάνω σχετικές τροπολογίες. Ε, η επιστημονική εξέλιξη του REACH ε, θα πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη την επαφή ε, και εδώ και το θέμα των κατευθυντήριων γραμμών και των νανοηλικών και τι γίνεται με κάποιες πρόσθετες ουσίες ή ακαθαρσίες που συμπεριλαμβάνονται. και τι γίνεται και με τις, ε, το RSFF ε, που είναι τροφές και ζωοτροφές. Και όπως είπε και η κυρία Σαλτεμόζε, θα πρέπει όλα αυτά να ενταχθούν στην κυκλική οικονομία. Δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί στα θέματα των ε, συσκευασιών και τι, στην έγχρωμη εκτύπωση, τι μελάνη χρησιμοποιείται, ακόμα αυτό δεν έχει λυθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. η κυρία Γιατερμάκη, επόμενη μιλήτρια είναι παρούσα μάλιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τις ε, ευχαριστίες και να ενώσω τη φωνή μου. Ήταν πολύ καλή συνεργασία πραγματικά με την κυρία Σάλντε Μόζε Όλοι οι σκιώδεις ηγητές είχαμε άψογη συνεργασία μαζί τους. Δεν ξέρω πολλά ζητήματα που είναι, τόσο ομόφωνη η Επιτροπή μας. Για την εναρμόνιση, για την ε, ε επαφή των τροφίμων με τα υλικά αυτά κτλ. Είναι περίπλοκη η κατάσταση και είναι πολλές ε, οι ουσίες που δεν γνωρίζουμε, που συμπεριλαμβάνονται στις συσκευασίε ή που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Δεν έχουμε πάντα και την ε, πληροφόρηση που χρειαζόμαστε για ε, το τι σημαίνει αυτό. Βέβαια τα επιστημονικά δεδομένα προοδεύουν και είναι σημαντικό να έχουμε γνώση των τελευταίων εξελίξεων όταν λαμβάνουμε αποφάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις και την αξιολόγηση που κάνουμε, πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η ενημέρωση αυτή δεν φτάνει ε, σε όλους τους ενεχομένους. Αυτό χωράει βελτίωση. Τώρα που ζητούμε περισσότερη εναρμόνιση για ένα κανονισμό, την ώρα που το ζητάμε αυτό θα πρέπει να έχουμε αρκετά επιστημονικά δεδομένα για να το τεκμηριώνουμε και να το στοιχειοθετούμε και από την άλλη θα πρέπει να έχουμε τους απαραίτητους πόρους για να ελέγχουμε την εκτέλεση και την εφαρμογή των κανονισμών αυτών. Τι νόημα έχει να έχεις κοινού ε, κανονισμούς αν δεν έχεις και τις ίδιες μεθόδους να τα ελέγχεις όλα αυτά. το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι οι ουσίες αυτές όταν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ε, μπορούν να έχουν ε, χημικά κατάλοιπα στα τρόφιμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και ένας άλλος ε, κίνδυνος από άλλα χημικά. Στο και τη σχετική νομοθεσία είναι πολλή δουλειά ακόμα που έχουμε. Πάντα όταν μιλάω για ουσίες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Δεν είναι εύκολο κάθε φορά να μετριέται η τοξικότητα των υλικών. Και όσο προχωρούμε προς μια κυκλική οικονομία, όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. θα πρέπει λοιπόν να μειωθεί η ε, ε, χρήση αυτών των τοξικών ουσιών. Αυτό που εγώ παγίως ζητώ είναι αυτορύθμιση, δηλαδή ε, εθελοντικές ε, ρυθμίσεις στη βιομηχανία. Η αυτορύθμιση λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. θα πρέπει η βιομηχανία να κανονίζει μόνη τη αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εκ. Ο κύριος Εκ. Α, δεν θέλω το λόγο, όχι. Προχωρούμε. Ο κύριος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σαλντεμόζε για την καλή προκατακτική δουλειά που έχει κάνει. Έκανε και ολόκληρη εκδήλωση. Είναι πολύ καλή η βάση, η έκθεσή της για την περαιτέρω συζήτηση και συμφωνούμε οπωσδήποτε κι εμείς ότι χρειάζεται καλύτερη εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χωρά καμία αμφιβολία και ούτε συζήτηση. Και η ΕΦΣΑ ε, πρέπει να ε, δουλεύει καλύτερα για να έχουμε καλύτερη βάση για απόφαση. Για να μην γίνονται παρεξηγήσει. Εμεί οι πράσινοι δεν έχουμε καμία μανία με την ΕΦΣΑ, αλλά να κάνει σωστά τη δουλειά τη. Βεβαίω υπάρχουν προβλήματα και δεν πρέπει να το ε, αποκρύπτουμε αυτό όταν κάνουμε εισαγωγέ από τρίτε χώρε. Θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια όπω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εσεί που προκαλούν ενδοκρινικέ διαταραχέ, οι περίφημοι ενδοκρινικοί διαταράκτες, που δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Είναι ένα πρόβλημα που μέχρι τώρα υποτιμάται, αλλά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλο και πιο σοβαρά. Και αυτό που χρειάζεται είναι όντως εναρμόνιση των διατάξεων. Ας πούμε για τα παιδικά παιχνίδια. Δεν μπορούμε από εκεί να απαγορεύουμε κάποιες ουσίες και να τις ε, βρίσκουμε μπροστά μας σε κάποιες συσκευασίες ενώ απαγορεύονται στα παιδικά παιχνίδια. Κάτι που μάλλον δεν ανέφερε πολύ η κυρία Σαλδεμόζα είναι το ζήτημα των ε, αποβλήτων. Όλοι φιλοδοξούμε να έχουμε μια κυκλική οικονομία και έχουμε αντικρουόμενα συμφέροντα από τη μια την προστασία των ε, τροφίμων και από την άλλη την ανακύκλωση. Αλλά το θέμα αυτό των αποβλήτων θα πρέπει να το λύσουμε με την ανακύκλωση όσο γίνεται περισσότερη ανακύκλωση για να μειωθούν τα απόβλητα. Άλλα θέματα που αναφέρθηκαν και προηγουμένως, τα νανοηλικά ε, τα ε, χρώματα που χρησιμοποιούνται στην εκτύπωση και το κοκτέιλ, δηλαδή ε, ουσιών ε, που αναμεγνύονται σε μία συσκευασία και τέλος καλύτερη συνεννόηση και καλύτερη πώς να το πω, καλύτερο συντονισμό της νομοθεσία αυτή με την νομοθεσία REACH. Εκεί υπάρχει έδαφος για βελτίωση και για εναρμόνιση. Αυτά νομίζω έχουμε μια πολύ καλή βάση για να κάνουμε καλή συζήτηση και τελικά καλή έκθεση. Ακόμα και αν πιέζει ο χρόνος, προλαβαίνουμε. Τουλάχιστον το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει μια καλή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. And the is Mr. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω, θέλω να κάνω ένα σύντομο σχόλιο σε σχέση με τα μόλις ακούσαμε. Όταν οι πράσινοι λένε ότι πρέπει να είμαστε πιο σταθεροί, πιο αποφασιστικοί για το θέμα των ενδοκρινικών διαταρακτών, ίσως θα μπορούσαν να υπογράψουν και την πρόταση μορφή που έχουμε κάνει για αυτό το θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πράσινοι είναι την Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και την κυρία Σαλδερμόζερ για την εργασία που έκανε. Ε, τα υλικά που βρίσκουμε στις συσκευασίε, ε, το χαρτί, ε, το πλαστικό ή στα διάφορα δοχεία όπως οι κατσαρόλες ε, μπορεί να μεταφέρουν χημικές ουσίες στα τρόφιμα και να τα μολύνουν. Είτε άθελα στη διάρκεια της κατανάλωσης, είτε είναι ουσίες οι οποίες έχουν προσθεθεί ακουσίως, όπως ας πούμε διάφορες ε, βρωμιές ε, καθαρσίες. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της, ε, δια, της, ε, διασύνδεσης των τροφίμων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και της ε, και κυκλικής οικονομίας. Επίσης, διατάξεις για τις χημικές ουσίες. Συμφωνούμε επίσης για την ανάγκη να εγγυηθούμε ότι οι νοσηρές ουσίες που κανονικά εξαλείφονται ε, με, βάση την οδηγία για τις χημικές ουσίες θα, διαγράφονται και από τη λίστα για τα ε, ουσίε που μπορούν να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Δηλαδή θεωρούμε πως θα πρέπει να γίνονται in vitro δοκιμές υποχρεωτικές ε, όσον αφορά την ανείχνευση των ενδοκρινικών διτρακτών μαζί με δοκιμέ για την νοσηρότητα. Τώρα όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου είναι σημαντικό να, να αντιπαραθέσουμε τα, τα στοιχεία για την τοξικότητα με, για τον άνθρωπο. Όχι μόνο δηλαδή τοξικότητα τη τροφίμου αλλά και την τοξικότητα τη επιφανία με την οποία έρχεται αυτό, το τρόφιμο σε επαφή. Υπάρχουν ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο κριτήρια μικροβιολογικά για την ασφάλεια σε σχέση με την αποδοχή των ε, διατροφικών προϊόντων και γι' αυτό θα ήθελα να δούμε αν και κατά πόσο θα πρέπει να εισαχθούν ε, ανάλογα κριτήρια για τα, ε, για τα υλικά τα επικίνδυνα που προορίζονται για να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και άρα να μεταφέρουν βακτήρια. Δεν συμφωνώ να αυξηθεί ο προπολογισμό του οργανισμού για την ασφάλεια των τροφίμων. Πολλέ φορέ την έχουμε επικρίνει ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο λειτουργία τη. Οι πολίτε θέλουν διαφάνεια, να ξέρουν αν πραγματικά λειτουργεί ε, για το δικό του συμφέρον και η ΕΦΣΑ από αυτή την άποψη είναι ανεπαρκή. Ευχαριστώ. Thank you. And next is Madame Merci, euh, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση συναδέλφου μας ε, ε, εντοπίζει πολύ συγκεκριμένα ζητήματα και πολύ σωστά τη συγχαίρω. Ε, είμαι πεπισμένη ότι η εναρμόνιση σε αυτόν τον τομέα είναι απολύτως απαραίτητη για την καλλιτουργία της εσωτερικής αγοράς και αποφεύγει στρεβλώσεις. Παρ' όλα αυτά η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει προς τα πάνω με πιο συγκεκριμένες προδιάγραφες και πρότυπα, πιο απαιτητικέ και με την ε, λογική της ε, σύνεσης. Μιλούμε για καθημερινούς κινδύνους, διότι η έκθεση σε ορισμένα υλικά είναι επαναλαμβανόμενη καθημερινή και από πολύ μικρή ηλικία. Καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί από ό,τι σε άλλα θέματα. Χαίρομαι που η έκθεση στηρίζει την έκθεση, την, ε, το ρόλο αξιολόγησης κινδύνου της ΕΦΣΑ. Όμως να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση αφορά την παράγραφο 6. Υπογραμμίζεται και πολύ σωστά το κόστος της αξιολόγησης κινδύνου. Και μετά καλείται να αυξηθεί ο προπολογισμό της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλείας Τροφίμων. Πράγματι, ε, χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική αρχή ασφάλειας τροφίμων που θα έχει τα κατάλληλα μέσα. Όμως, λέτε ότι υπάρχουν εθνικά περιθώρια για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού. Όμως, όσο η διαδικασία εναρμόνισης δεν έχει ολοκληρωθεί, μπορούμε να πούμε ότι οι αποφάσεις, οι εθνικές αποφάσεις ε, ή οι ε, ε, εθνικές αρχές τροφίμων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα άλλο σημείο για την αξιολόγηση κινδύνου είναι το εξής. Τα κριτήρια ε, ορισμού των ενδοκρινικών διαταρακτών στη, στα προϊόντα ε, ή στα υλικά, τα επιβλαβή υλικά. Πράγματι, επανερχόμαστε πολύ συχνά σε αυτό το θέμα. Όμως για ποιο λόγο. Γιατί ε, είναι πολλά τα συμφέροντα ε, και πολλά τα προβλήματα. Θα πρέπει να πάμε πιο μακριά. Να καθορίσουμε συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης ε, ταξινόμησης και να ενισχύσουμε τα υγειονομικά μέτρα που λαμβάνουμε προκειμένου να λάβουμε υπόψη τους ενδοκρινικούς διαταράκτες που γενικά επηρεάζουν και θα επηρεάσουν πολύ βαθιά την υγεία των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. Thank you. This was uh, the end of our... Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ ο πρώτος γύρος. Και έχουμε και δεύτερο γύρο. Τώρα από τα μέλη της Επιτροπής μας, αφού ακούσαμε τους Σκιώδης, η κυρία Μπόιλαν, ευχαριστώ ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ και για τη συζήτηση. Ε, αυτό το θέμα πραγματικά δεν έχει συγκεντρώσει ε, τη δέουσα προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης ακούμε τους συναδέλφους ε, και βλέπουμε ότι συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ε, ρύθμιση για αυτές τις ουσίες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Που είναι 15.000 και πλέον οι ουσίες που χρησιμοποιούνται ε, στις συσκευασίε και τα τρόφιμα είναι από τις βασικές πηγές της έκθεσης του ανθρωπίνου οργανισμού σε χημικά. Υπάρχουν επικίνδυνα υλικά Ε, και ε, προφανώ υπάρχει το επιχείρημα ε, ότι στι συσκευασίε που έρχονται επαφή με τρόφιμα είναι μεγαλύτερη προσοχή που δίνουν. Αλλά ακούμε ότι 13 από τα 17 μέτρα δεν είναι εναρμονισμένα όπως ακούσαμε. Είναι πολύ εμβαλωματικές οι λύσεις και η προτινόμενη νομοθεσία μπορεί να είναι κάτι καλό, αλλά δεν εφαρμόζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα πρέπει λοιπόν από τις ε, ε, συσκευασίες αυτές να περνούν στα τρόφιμα ουσίες που είναι ε, επικίνδυνες για τον ανθρώπινο οργανισμό ή επιβλαβής. Μια πρόσφατη μελέτη της ΕΦΣΑ λέει ότι, ότι είναι ενεαπλάσια ε, η, έκθεση ε, τέτοιων συσκευασιών Μάλλον συγκέντρωση ε, σε επικίνδυνες ουσίες για τρόφιμα ή προϊόντα που προορίζονται για νεογνά ή για βρέφη. Και έχουν πλέον και τα τρόφιμα αυτά ε, μακρύτερη διάρκεια ε, ζωής και παραμονή στα ράφια των ε, καταστημάτων που σημαίνει ότι έρχονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τα τρόφιμα σε επαφή με τις συσκευασίε. Και μπορεί και ακόμα και μικρή δόση να έχει τεράστιο τεράστια, πώς να το επίδραση και να προκαλέσει βλάβη σε ένα βρέφος, σε ένα νέο γνώ. Είναι απαράδεκτος λοιπόν ο κίνδυνος, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα βρέφη, επαναλαμβάνω, και τα ε, πολύ μικρά παιδιά. Θα ήθελα το σχόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έχει γίνει μια μελέτη ε, ε την οποία κρατά μυστική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν τη δημοσίευε. Για ποιο λόγο τα κριτήρια EDC ήδη έχουν καθυστερήσει. Θα ήθελα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη ρωτήσω και να τη ζητήσω να μας πει γιατί δεν τα δημοσιεύουν αυτά τα στοιχεία, κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι ε, απαραίτητο απαραίτητο να ενισχύσουμε την αρμόνιση όλων αυτών των υλικών. Ορισμένε από τι χημικέ ε, αυτέ ενώσει που περιλαμβάνονται στα υλικά έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και αυτό ενισχύει του πολίτε μα και του θέτει σε κίνδυνο. Συγχαίρω την εισηγήτρια. Ε, είναι κρίμα που έχουμε ένα ολόκληρο κατάλογο 17 υλικών και από αυτά τα 17 μόνο 4 έχουν τύχη εναρμόνισης μέσω ειδικών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι τρομακτικό γνωρίζοντας ότι ε, όλα αυτά τα υλικά περιέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Μιλάμε για χαρτιά, για χαρτί, για χαρτόνι. Εγώ θα σας μιλήσω για πλαστικό και θα συνδέσω το θέμα αυτό με το θέμα των ενδοκρινικών διατρακτών. Γνωρίζω ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ταμπού, αλλά για αυτό το λόγο επιμένω, διότι ε, θέλουμε η, η χημική σύνθεση των πλαστικών που έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα να ελέγχεται. Απαραίτητο, αλλά πώς θα πετύχουμε αυτό το στόχο χωρίς ειδικό κανόνα που να αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Μια και αυτοί είναι παρόντες στην πλειοψηφία αυτών των προϊόντων. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία τον ορισμό που μας έχει υποσχεθεί πριν το καλοκαίρι η Κομισιόν. Παράδειγμα, παράγραφος 10 της έκθεσης της ε, κυρίας Σαλδεμούς που δικαιολογεί την μείωση του ορίου μετανάστευσης της, της διφενόλης α ε, που περιλαμβάνεται στα, ε, στις συσκευασίε και στα πλαστικά. Ε, όμως υπογραμμίζει ταυτόχρονα ότι αυτό το όριο μετανάστευσης, αυτό το ανώτατο δεν εφαρμόζεται σε όλα τα υλικά τα οποία έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Γνωρίζουμε του σοβαρού κίνδυνους από την άλλη μεριά που συνδέονται με τη διφενόλη Α ω ενδοκρινικό διαταρακτή. Σα υπενθυμίζω ότι στη Γαλλία απαγορεύεται σε όλους τους σε ε, περιεκτές τροφίμων από το 2015, από τον Γενάριο του 2015. Συνεπώς υπάρχει μια έλλειψη συνέπειας, ε, μια λογική ασυνέπεια, διότι ε, θέλουμε να χειριστούμε όλα αυτά τα υλικά, χωρίς όμως να καθορίζουμε συγκεκριμένους κανόνες για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Υποστηρίζω λοιπόν την έκκληση της εισηγήτριας να αναθεωρήσουμε το σημερινό ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά ειλικρινά αυτό θα πρέπει να γίνει υπό το φως καινούριων κανόνων που θα υιοθετήσουμε για τις ε, ουσίες που δρούν και επηρεάζουν το ενδοκρινικό σύστημα. Κύριε Μελχιόρ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σήμερα συζητούμε για τις ουσίες αυτές που περιβάλλουν τα τρόφιμά μας και μεταδίδονται δεχομένως και στα τρόφιμα. Και χρειάζεται ακριβώς να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, να αφιερώσουμε χρόνο για ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ την συγγήτρια Κρίστελ Σαλντεμόζε από καρδιάς για την έκθεσή της. Ε, τα σημαντικότερα σημεία περιλαμβάνονται σε αυτή ήδη. Μπορώ να συμφωνήσω και να υπογραμμίσω τα όσα είπαν οι προλύσαντες συνάδελφοι. Ανησυχούμε κι εμείς ότι από τις 17 ουσίες δεν έχουν εναρμονιστεί όλες και ενώ υπάρχει ενιαία αγορά υπάρχει πρόβλημα για τους ελέγχους. Αν δεν έχουμε εναρμονισμένους κανόνες πώς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ουσιαστικό έλεγχο. Και ιδιαίτερα Ακριβώς επειδή δεν είναι δεδομένη η αμοιβή αναγνώριση, αν ήταν θα υπήρχε δυνατότητα και ελέγχων. Όλα αυτά δεν λειτουργούν. Ε, με βάση όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ε, είναι απολύτως και επιγόντως απαραίτητη η εναρμόνιση αυτή και κάτι άλλο που πιστεύω και ε, αναφέρθηκε επανειλημμένα από τη μια έχουμε την ΕΦΣΑ, από την άλλη έχουμε και το ΡΙΤΣ τον οργανισμό για τα χημικά που θα πρέπει να αποφαίνεται για κάποιες ουσίες και να ορίζει κατά πόσο ε, ενδέκνεται ή όχι, είναι κατάλληλες ή ακατάλληλες για επαφή με τρόφιμα. Για να γίνουν όλα αυτά, ε, χρειάζεται συνεργασία αυτών των οργανισμών. Δεν μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα έτσι. Ε, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το προωθήσουμε αυτό. Αφήστε δε που είναι και το ταμείο μία. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια και είμαι βέβαιη ότι θα καταλήξουμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα πολύ καλό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιέλνερ. πολύ καλή έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό για την εσωτερική αγορά να διαθέτουμε ομοιόμορφους κανόνες για αυτά τα υλικά και όπως ακούσαμε μόνο τέσσερα από τα 17 υλικά τα οποία έχουν ε, περιληφθεί στον κατάλογο ε, έχουν τυχαία εναρμόνισης. Χωρίς να πω σε λεπτομέρειες όμως, να πω το εξής. Είναι πολύ σημαντικό το χαρτί και το χαρτόνι τουλάχιστον να ε, συμπεριληφθούν ε, στα εναρμονισμένα υλικά. Διότι και εκεί θα πρέπει να γίνει διαφορά, διάκριση ανάμεσα στα καινούργια και τα ανακυκλωμένα υλικά. Κάποιοι θα πούν δεν πρέπει να κάνουμε διακρίση, γιατί θα πρέπει να προωθήσουμε την κυκλική οικονομία. Όμω, μπορούν να γίνουν και τα δύο. Γιατί έχουν διαφορετικέ ιδιότητε τα καινούργια από τα ανακυκλωμένα. Οπότε θα πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Δεύτερον, ε, έχω κάποια προβλήματα σε σχέση με το πώς συζητάμε το, ε, το φαινόμενο κοκτέιλ. Αυτό αποκαλούμενο φαινόμενο κοκτέιλ. Η ΕΦΣΑ έχει να παίξει, έχει να παίξει ρόλο και θα πρέπει να λάβει υπόψη τα περιθώρια ασφαλεία τα οποία αφορούν το, το φαινόμενο κοκτέιλ. Όμω, το φαινόμενο κοκτέιλ ω όρο χρησιμοποιείται με διαφορετικού τρόπου από διαφορετικού ανθρώπου. Δεν υπάρχει σαφής ορισμό αυτή τη στιγμή. Αν όμω πούμε ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία αυτή για να λάβουμε υπόψη γνωστές ουσίες που έχουν γνωστές συνέπειες, αυτό γίνεται ήδη. Γίνεται να γίνει. Μπορεί να γίνει, αλλά με την αρχή της προφύλαξης, την οποία ήδη χρησιμοποιεί βέβαια. Με ε, τιμές ασφαλείας και περιθώρια ασφαλείας. Μεγάλα περιθώρια ασφαλείας όμως. Μερικές φορές αυτά φτάνουν και στο 100% για να ληφθούν υπόψη τέτοιου είδους ε, φαινόμενα όπως το φαινόμενο κοκτέιλ. Αν όμως εννοούμε κάτι διαφορετικό και όχι γνωστές ουσίες με γνωστά αποτελέσματα θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα τον όρο. Τέλος, να πω το εξή. Οι ποιότητες νομοθεσία είναι ένα πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η εφαρμογή και ένα τρίτο πρόβλημα είναι τα κράτη-μέλη να σέβονται την νομοθεσία. Γιατί η διφενόλη, για παράδειγμα, ε, για τη διφενόλη υπάρχουν καινούργια κατόφλια από την ΕΦΣΑ, αλλά τελικά τα κράτη-μέλη κάνουν ό,τι θέλουν. Η Γαλλία, για παράδειγμα, μέσω της εθνικής της νομοθεσίας, πολύ πρόσφατα, ε, που υιοθέτησε πολύ πρόσφατα, παραβιάζει τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς η Κομισιόν θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα κατόφλια και οι κανόνες που παράγει η ΕΦΣΑ ε, τη χάνουν σεβασμού. Γιατί αλλιώς δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε νομική ασφάλεια στην εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και αυτό. Ακόμα και εκεί που ήδη έχουμε ήδη κατόφλια. Η Κομισιόν ε, δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου. Ευχαριστώ. Ωραία, θα πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση εδώ. Θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει στις ε, παρατηρήσεις που έγιναν από την εισηγήτρια, τους και εισηγητές και τα μέλη της Επιτροπής. Έχουμε άλλο ένα θέμα στην μεσαία διάταξη. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να μην μακρηγορήσει. Τρία-τέσσερα λεπτά μόνο παρακαλώ. Κυρία Γκλέσιας. thank you. Thank you very much. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρωτοβουλία αυτή που αναλάβατε να αναθέσετε την συγκεκριμένη μελέτη αξιολόγησης προκειμένου να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης. Όπως γνωρίζετε η Κομισιόν ολοκληρώνει σύντομα μια μελέτη που εξετάζει την κατάσταση ό,τι αφορά τα εθνικά μέτρα και την χρήση των υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και τα οποία δεν έχουν εναρμονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης εξετάζουμε την κατάσταση των εναρμονισμένων υλικών και το πώς λειτουργεί αυτή η εναρμόνιση σε εθνικό επίπεδο. Όταν συλλέξουμε όλες αυτές τις πληροφορίες μαζί και την μελέτη που μας παρουσιάσατε σήμερα, θα έχουμε πλέον μια καλύτερη εικόνα των προβλημάτων και κατά αυτόν τον τρόπο θα εξετάσουμε αν πρέπει να αναλάβουμε δράση σε ό,τι αφορά τα υλικά σε επαφή, που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα στο μέλλον η βιομηχανία μας έχει ζητήσει επανειλημμένως ε, να υιοθετήσουμε καινούριου κανόνες για να διευκολύνουμε την εσωτερική αγορά. Όπως γνωρίζετε όμως, ε, η νομοθεσία θα πρέπει να είναι ανάλογη με το, τους στόχους και να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας. Η παρούσα κατάσταση είναι τεχνικά περίπλοκη. Το απέδειξε αυτό η σημερινή συζήτηση. Συνεπώς, δεν θα είναι ε, η λύση δεν θα είναι απλή και εύκολη. Η περίπτωση των πλαστικών είναι ε, πολύ γλαφυρή. Πριν γίνει οποιαδήποτε λεπτομερή εναρμόνιση άλλων υλικών, πριν απαιτήσουμε συγκεκριμένες δράσεις από τη βιομηχανία και ε, πριν αναλάβει δράση η ΕΦΣΑ, είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε, να αξιολογήσουμε αν τέτοιου είδου διαδικασίες είναι απαραίτητε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εναλλακτικέ λύσεις έναντι αυτού του συστήματος θα μπορούσαν επίσης να εξερευνηθούν για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των τροφίμων και την, ε, το σεβασμό των αρχών της εσωτερικής αγοράς. Δεν πρόκειται να απαντήσω σήμερα στην ερώτηση των ενδοκρινικών διαταρακτών, αλλά όπως σας είπα η Κομισιόν εργάζεται προκειμένου να βρει την καλύτερη λύση. Για αυτό το θέμα το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά. Ευχαριστώ. Hey, Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να απαντήσει πάρα πολύ σύντομα μέσα σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εισηγήτρια. Ε, όλους τους συναδέλφους για τα εξαιρετικά τους ε, σχόλια. Ιδιαίτερα όταν είπατε ότι χρειάζεται περισσότερη εναρμόνιση και ειδική αντιμετώπιση για όλες τις ουσίες, όντως. οι χημικές ουσίες και οι ενδοκρινικοί διακτάρακτες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω να έχουμε μεγάλη πλειοψηφία στην ψηφοφορία και στις τροπολογίε. Ευχαριστώ ε, και την συγκεκριμένη και τους κοιόδης. Προθεσμία τώρα κατάθεση τροπολογιών ε, είναι η Δευτέρα Ιουνίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 11 και 12 Ιουλίου και στην Ολομέλεια Οκτώβριο. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας στη συζήτηση αυτή. Προχωρούμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα στη μέση διάταξη. Ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 106, διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρίφαλου. Παρακαλώ. Ε, συνεισηγητές Αρχίζουμε τη συζήτηση, δηλαδή τι αρχίζουμε, έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Και κανονικά σε 10 λεπτά τελειώνει και η διερμηνία. Θα σας παρακαλούσα να περιοριστείτε σε 2 λεπτά. Ο κύριος Μπάρτ Στάς έχει το λόγο. Τώρα που έχουμε ακόμα διερμηνία να τα πω ολλανδικά. Είναι η νιωστή ένσταση ε, την οποία κάνουμε με τους συναδέλφους Μπαλάς, Εύη, ε, Μπόιλεν και Πιέτικάινεν, αυτή τη φορά πρόκειται για ένα λουλούδι, το γαρίφαλο, ε, γεννητικά τροποποιημένο και για αραβόσιτο. Τα δύο θέματα διαφέρουν. Για το γαρίφαλο υπάρχει ειδική παρατήρηση ότι μόνο 11 κράτη-μέλη ήταν υπέρ 36% του πληθυσμού. Η Εύσα τι λέει. Από ό,τι φαίνεται γνωρίζει η Εύσα ότι τα φύλλα, τα πέταλα του γαριφάλου ε, ε, σε κάποιους ε, πολιτισμούς, σε κάποιες χώρες τα τρώει ο κόσμος, είναι τρόφιμο. και δεν ξέρουμε κατά πόσο ένα μεταλλαγμένο γαρίφαλο μπορεί να καταναλωθεί σκεμμένα ή τυχαία. Μπήκα στο ίντερνετ και βρήκα ένα σωρό συνταγές που έχει μέσα ε, γαρίφαλο. Γαρίφαλο το λουλούδι δηλαδή, όχι το μπαχαρικό. Και λέει η Εύσα ότι η γύρι από αυτά τα μεταλλαγμένα ε, μπορεί να μεταδοθεί και υπάρχει κίνδυνος ε, ε, επιμόλυνσης των καλλιεργειών. Εν πάση περιπτώσει έχουμε την ένσταση αυτή δεν έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη θέματα δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος. Έρχομαι τώρα στον Αραβόστο. Είναι περίπου η ίδια επιχειρηματολογία ε, και σε σχέση με την προηγούμενη έσταση. Τώρα μετά το νέο πλαίσιο που έχουμε και μετά το γεγονός ότι η μόνιμη επιτροπή για τα φυτά και την ασφάλεια ε, συνεδρίασε την περασμένη φορά. Αυτό το καλαμπόκι ε, Αθίσταται στο γλυφοσάτ και σε αυτή την πολιτική συγκυρία που ζούμε, που δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν για την ε, παράταση της άδεια κυκλοφορίας στο γλυφοσάτ στην αγορά, ε, δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια φαινόμενα να εγκριθεί αυτό το καλαμπόκι. Ε, σταματώ προς το παρόν εδώ. Ευχαριστώ κύριος Μπαλάς. Μάλιστα, θα είμαι σύντομο γιατί τα βασικά τα είπε ο συνάδελφος Μπαρτεστές, Δεν έχω πολλά να προσθέσω για το πρώτο σημείο να πω ότι το πρόβλημα είναι πάντοτε το ίδιο. Το θέμα της ε, διάδοσης, ε, της, μάλλον της ε, ε, εξάπλωσης ε, του εισγύρης ε, που ανησυχεί και τα, περιπλέκει τα πράγματα. Το δεύτερο σημείο, το θέμα του αδραβόσιτου, για αυτή την υπόθεση της γλυφοζάτης είμαστε ενώπιον ενό ιδιαίτερου πράγματος, γιατί ψηφίσαμε κάτι εμείς εδώ το Ευρωκοινοβούλιο και έγινε και συζήτηση σήμερα με την όσον αφορά τον χρόνο που παραμένει ακόμα σε πώληση γλυφοσάτη. Πάντως στόχος είναι να μην πωλείται πλέον. Πώς μπορούμε να σκεφτούμε ότι σε 7-10 χρόνια θα μπορούμε να πάμε παντού, να βγάλουμε το, τον αραβόστο που είναι, αντιστέκεται στη γλυφοσάτη, γιατί η γλυφοσάτη δεν θα πωλείται πια και θα ληφθούν αποφάσεις και η υπόλοιπη επιχειρηματολογία έγινε για τις υπόλοιπες αντιρρήσεις. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Thank you, Boylan. Ευχαριστώ κύριε Μπόιλαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα κι εγώ να χαιρετήσω ε, την υποβολή αυτών των εστάσεων. Έχουν υπογράψει τα περισσότερα μέλη των πολιτικών ομάδων και βλέπετε ότι αυτό είναι διακομματικό δεν είναι θέμα κομματικό, γιατί υπάρχουν ελλείψεις στον τρόπο με τον οποίο εκρίνονται τα μεταλλαγμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη φορά ε, είναι η έκτη ένσταση, η συγκεκριμένη μάλιστα η πέμπτη και η έκτη, ε, που είμαστε απέναντι στα γενετικά τροποποιημένα. Είπαν οι συνάδελφοι πρόκειται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω αν μας ακούει ή αν σοβαρά προσπαθεί ε, να αντιμετωπίσει το θέμα. Έχει περάσει ένας χρόνος και παραπάνω από τότε που έκανε αυτή την πρόταση και οι ευρωβουλευτές το απέρριψαν. Και εξακολουθούν να θέλουν να περάσουν με τη βία εγκρίσει και άδειε χωρίς να υπάρχει ειδική πλειοψηφία ε, από τα κράτη-μέλη με την καταγραφή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποτίθεται ότι είναι και δημοκρατική η λήψη των αποφάσεων εδώ πέρα μέσα. Η ένσταση την οποία συζητούμε σήμερα αφορά ε, αυτό το γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι που ανθίσταται στην Και ε, Είδαμε πόσο έολο είναι το σύστημα έγκρισης διαδιοδότησης ε, για τα μεταλλαγμένα. Εύσα γνωμοδοτεί και θα πρέπει να βασιστεί για την απόφαση να βασίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν ανταποκρίνεται ε, στο έργο της. Ε, οι πολίτες ανησυχούν, είναι και καρκινογόν αυτά τα πράγματα. Οπότε, όπως Γίνεται λόγο στο εμπορικό απόρριτο. Είναι, λέει, αρκετό λόγο για να μην μα ε, κοινοποιούν τα στοιχεία ακόμα και αν πρόκειται για το δημόσιο συμφέρον. Υπάρχει όμως η διαδικασία αυτή σχετική με τη γλυφωσάτη και το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ κυρία Εύη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πέρα από τις ε, αιτιολογήσεις που υπέβαλαν οι παρουσίασαν μάλλον οι συνάδελφοι με τους οποίους έχω συνυπογράψει την ένσταση, εγώ θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα που αφορά μια πτυχή που ήδη ενεφέρθηκε δηλαδή το πόσο είναι δημοκρατική αυτή η διαδικασία έγκρισης των, ε, μετα, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Σήμερα, μέχρι σήμερα δεν είναι ε, και θα πρέπει να δούμε τι κάνουν οι τεχνικές επιτροπές όταν, ας πούμε, σε περίπτωση μη έκδοση γνωμοδότηση από αυτές τις επιτροπές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτόνομα εγκρίνει. Αδειοδοτεί. Θα ήθελα να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι για την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού 715 του 2005 σε σχέση με τις εκπομπές ε, των ε, αυτοκινήτων. Έχω μια πρόταση επιτάπητος που λέει ότι ε, σε περίπτωση που δεν εκδώσουν νομοδότηση οι αρμόδιες επιτροπές, η, Επιτροπή, η Κομισιόν δεν θα μπορεί να εγκρίνει και την κυκλοφορία στην αγορά του τάδε του δίνα, οποιαδήποτε δηλαδή ε, ουσίας. Δεν μπορεί η Κομισιόν να αδειοδοτεί γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς χωρίς να υπάρχει δημοκρατική διαδικασία που να ακούει την γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ και τώρα οι δύο ομάδες που δεν υπέγραψαν την ένσταση. Πρώτα Φιέλνερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχά είναι να ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό δεν, πρέπει να, δεν είναι μια διαδικασία για το κατά πόσο μα αρέσει ή όχι. Είναι μια διαδικασία που σαφώ ορίζεται ως ένα εργαλείο για το Κοινοβούλιο, ώστε το Κοινοβούλιο μάλλον να μπορεί να ελέγχει και να ενεργεί, εφόσον η Κομισιόν δεν ακολουθεί την νομοθεσία που εμείς έχουμε ε, συστήσει, όσο σκληρή και αν είναι αυτή, ή εάν η Κομισιόν παραβλέπει τις επιστημονικές αποδείξεις. Αυτά είναι τα κριτήρια. Δεν πρόκειται για την κλειφωσάτη. είναι ε, το θέμα κατά πόσο η Κομισιόν ε, ακολουθεί τους κανόνες. Ε, η Κομισιόν έχει ξεπεράσει την εντολή της. Εγώ δεν άκουσα ούτε ένα επιχείρημα. Κανένας δεν προσπάθησε καν να το αποδείξει αυτό. Δεύτερον, η Κομισιόν έχει παραβλέψει επιστημονικές αποδείξεις. Όχι, θα έλεγα εγώ. Έχουμε ζητήσει την ΕΦΣΑ να είναι το επιστημονικό μας σώμα. Η ΕΦΣΑ για τα γαρίφαλα στην SHD 25531 Παύλα 4 κατέληξε ότι η ε, πορεία του γενετικά τροποποιημένου γαρίφαλου δεν θα προκαλέσει ε, αρνητικέ επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον. Η ίδια απόφαση ε, λήφθη στις 7 Δεκεμβρίου, αλλά δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Και με όλο τον σεβασμό στον κύριο Στάς, Γκουγκλάροντας για άλλα παραδείγματα, εάν ζητήσουμε από ένα συγκεκριμένο σώμα να είναι ο επιστημονικός μας σύμβουλος, θα πρέπει να σεβαστούμε τις αποφάσεις του. Εμείς ζητήσαμε από την ΕΦΣΑ να κάνει τη δουλειά αυτή. Μας έδωσε ένα συγκεκριμένο πόρισμα που δεν μας αρέσει όμως. Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν είναι βάσιμα, δεν, δεν στέκουν. Κατανοώ και μάλλον κατανοώ ότι πολλοί συνάδελφοι δεν συμπαθούν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και είχαμε καταψηφίσει και την τελευταία φορά τον κανονισμό γιατί δεν θέλαν. Εγώ το έκανα για διαφορετικό λόγο, αλλά δεν ψηφίσαμε μορατόριο. Το απορρίψαμε για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δεν ξέρω τι προσπαθείτε να μας κουράσετε με αυτές τις συζητήσεις και να σταματήσετε τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς με αυτόν τον τρόπο. Πάντως είναι ο λάθος τρόπος. Λάθος τρόπος για νομοθεσία. Ευχαριστώ. μάνα. Ευχαριστώ πολύ. Στην Άλντα είχαμε τη συζήτηση αυτή κι εμείς και προσπαθήσαμε να το δούμε με τρόπο ρεαλιστικό και πραγματικά. Δύο είναι οι λόγοι κάθε φορά για τις εντάσεις αυτές. Πρώτος λόγος είναι να ε, κουραστεί πραγματικά και να ε, καταρρεύσει όλη αυτή η διαδικασία για την ε, διοδότηση και να μπορούν τα κράτη-μέλη να ε, απορρίπτουν πιο εύκολα ε, τα γενετικά τροποποιημένα. Αυτό εκνεύρισε, εξόρισε κάποιους συναδέλφους και θέλουν να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς αυτά δεν τα μασάμε και δεν πρόκειται να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερον, ορισμένοι δεν θέλουν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς γενικώς. Ακόμα και αν δείξει ε, η επιστημονική έρευνα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα ζώα, για το περιβάλλον και σε καμία περίπτωση ε, για την ανθρώπινη δημόσια υγεία, παρόλα αυτά σου λέει όχι. Γι' αυτό ζητήσαμε να ε, τα κοιτάξει που είναι ένα ανεξάρτητο επιστημονικό όργανο, ό,τι υπάρχει στον κόσμο, ό,τι κυκλοφορεί, να δει τι ευσταθεί και τι δεν ευσταθεί. Ε, είναι επιστημονικά στοιχεία και τώρα έχουμε βουλευτές που ψάχνουν στο Google νέες μελέτες και το ξανανοίγουν πολιτικά. Δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να εμπιστευτούμε την ΕΦΣΑ. Εμείς τους δώσαμε αυτή την ε, ε, εντολή και για το γλυφοσάτι και πάλι συνδέεται με τις γενετικά τροποποιημένους. Ε, είναι μεταλλαγμένα, είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Ε, γιατί θέλετε να απαγορευτεί η γλυφοσάτη, είναι από τα πιο ε, ανώδυνα προϊόντα, από τα πιο ακίνδυνα. Υπάρχει εκεί και η αρχή της προφύλαξης. Δεν θέλετε δηλαδή ζυζανιοκτώνα καθόλου. Τα ζυζάνια να τα αφήνουμε, ε, να χρησιμοποιούμε πιο δυνατά φάρμακα ή με την άρρωση. Αλλά εάν κάθε φορά ε, πηγαίνουμε και οργώνουμε τα χωράφια, θα τα ρημάξουμε, θα αυξηθεί η διάβρωση, θα αυξηθεί η εκπομπή διοξίδιο ε, του άνθρακα, θα έχουμε περισσότερη διαρροή θρεπτικών ουσιών από το χώμα και δεν βοηθάει ούτε αυτό. Θα δώσω, θα δώσω το λόγο στην ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά τα σχόλια. Να σας καθυσυχάσω καταρχήν. Η Κομισιόν δεν έχει υπερβεί τις ε, αφραμοστικές αρμοδιότητες που τις έχουν δοθεί. Σας βεβαιώνω. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να αποσύρουμε την πρόταση. το δικαίωμα ελέγχου του Κοινοβουλίου αφορά μόνο το αν έχουμε υπερβεί τις αρμοδιότητες που μας έχουν χορηγηθεί και δεν τις έχουμε υπερβεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο κάποιων από τα σχόλια. Πρώτον, για το γαρίφαλο. Ε, πρόκειται για ε, ε, κομμένα λουλούδια παρόλα αυτά είναι γενετικό τροποποιημένο. Η ΕΦΣΑ συμπέρανε ότι δεν υπάρχει κανένα είδου επιστημονικό λόγος να μα ανησυχεί η ανθρώπινη υγεία ακόμα και αν κάποιο το καταπιεί, το φάει ή ακόμα και αν ε, η γύρι ε, ε, διαδοθεί, αποδράσει το περιβάλλον. Δεν υπάρχει πρόβλημα για το περιβάλλον. Ο, ο μάρκερ που χρησιμοποιείται ε, ε, δεν μπορεί να ε, βοηθήσει στην ανεφορίων ανάπτυξη του φυτού και δεν μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Η άδεια, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και υποχρεωτική σήμανση ότι πρόκειται για γενετικά τροποποιημένο γαρίφαλο και ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, για ανθρώπινη κατανάλωση, για κατανάλωση από ζώα και δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Οι δείκτες ε, που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι πιο αυστηροί ε, και μάλιστα το δικό μας σύστημα είναι το πιο αυστηρό σύστημα στον κόσμο. Σε ό,τι αφορά την, το γλυφοσάτ ε, και την ε, ανοχή στον ανθρώπινο οργανισμό. η, ο κανονισμός για τα παρασιτοκτόνα καθορίζει τα όρια και το πώς δίνονται οι άδειες. Από και εκεί είναι οι κανόνες. Ορισμένα μέλη αναφέρθηκαν και σε δημοκρατικό έλλειμμα. Η πρόταση που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2015 ανέφερε ότι μπορούν να γίνουν αλλαγές και έγιναν προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο στα κράτη-μέλη να λαμβάνουν υπόψη το ακριβές ε, εθνικό περιβάλλον. Οπότε προφανώς Λυπούμαστε που, αποσύρθηκε, που απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Δυστυχώς η διερμηνία θα πρέπει να διακοπεί αυτή τη στιγμή ε, και η συνεδρία θα συνεχιστεί στα αγγλικά. Into account. And as for any legislative proposal, the rules which are in place have to continue to be um, implemented uh, even during the negotiations.